Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε σήμερα δύο σύντομες ανταλλαγές απόψεων. Σήμερα όμως έχουμε 19 γλώσσες που διερμηνεύονται. Είμαστε πάντα στο διαδίκτυο και είμαστε και άχαρτοι, paperless, τα πρακτικά της 18ης ε, Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα και εάν δεν υπάρξουν σχόλια θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί και θέλω να συγχαρώ τον Ζεμ για, το, για τα γενέθλιά του σήμερα. θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Σούτσα και τον κύριο Μάρτιν για την πρώτη ακρόαση. Σας είπατε έχουμε δύο σύντομε ακροασει οπότε θα υπάρξει μονάχα ένας γύρος ερωτήσεων και όπως πάντα θα δώσω άμεσα το λόγο στον κύριο Σούτσα για να κάνουμε μερικέ ε, αρχικές ε, παρατηρήσεις και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. κύριε και κύριοι καλημέρα σα, <clears throat> σα ευχαριστώ που με ξανακαλέσατε. Λυπάμαι που η πρώτη μου παρουσία το Μάρτιο δεν μπόρεσε να γίνει δυνατή και χρειάστηκε να με αντικαταστήσει η Ταλίλα Καουντορή αλλά μπορέσαμε να σας δούμε στην επίσκεψή σας τον Ιούλιο στην Ίσπρα, η οποία ήταν πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, <clears throat> στο φως αυτών που συζητήσαμε τον Απρίλιο, αυτών που συζητήσαμε σε βάθος με την παρουσία σας δύο μέρες στην Ίσπρα, θα ήθελα να εστιάσω σε τρία σημεία στην εισαγωγική μου ομιλία και μεταξύ των τριών αυτών θα σταθώ περισσότερο στο τρίτο σημείο γιατί είναι σημαντικό να ατενίσουμε το μέλλον. Όχι μονάχα να αντλήσουμε συμπεράσματα από αυτά που έχουν γίνει, αλλά είναι απαραίτητο να δούμε ποιο είναι και το μέλλον. Πρώτα απ' όλα το Κοινό Κέντρο Ερευνών και η θέση του μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εναντί των κρατών μέλλων. Ξέρετε ότι είμαστε μια επιστημονική υπηρεσία της Κομισιόν και η εντολή μας είναι να υποστηρίξουμε σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο τη λήψη αποφάσεων στην Κομισιό, την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων, το, το 30% λοιπόν είναι σε, στο να βοηθούμε την προετοιμασία νομοθετημάτων και μετά έχουμε ένα 70% που υποστηρίζει την ε, εφαρμογή αυτών των νομοθεσμάτων στην πράξη. Έχουμε λοιπόν ε, ρόλο και στην κοινή αγροτική πολιτική και επίσης για την ε, ε, εκπλήρωση των προαπαιτουμένων σε ό,τι αφορά την βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα και επίσης σε ό,τι αφορά ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίμαχο, το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τίποτα δεν μπορεί να τεθεί στην αγορά εάν η Κομισιόν και το Κοινό Κέντρο Ερευνών δεν επικυρώσουν την αρμόδια μεθοδολογία. Αυτό λοιπόν είναι και η, κατάσταση στους τομείς που έχει εντολή η Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Μας δίδει την ε, σκητάλη σε τεχνικό επίπεδο, σε άλλα έχουμε ένα συμβουλευτικό και μόνο ρόλο. Σε λίγο θα είναι τα 60 χρόνια της δημιουργίας του Κοινού Κέντρου Ερευνών το 2017. δεκαετία του 80 ε, διευρύναμε τις δραστηριότητές μας από μονάχα τα θέματα ποινικής ασφάλειας σε θέματα ευρύτερα. Είμαστε ανεξάρτητοι, δεν δεσμευόμαστε από τη θέση της βιομηχανίας ή της κοινωνίας των πολιτών και ο στόχος μας είναι μέσα στην Κομισιόν να μπορέσουμε να οργανώνουμε συζητήσεις, έρευνες και να δίδουμε στοιχεία που να βασίζονται σε εμπεριστατωμένη γνώση. Αυτό ισχύει λοιπόν και για τις ε, εκπομπές από αυτοκίνητα οχήματα. Ξέρετε ότι υπήρχε το 2001 απόφαση της Κομισιόν του Επιτρόπου Μπουσπίσκια, ο οποίος θεώρησε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα των εκπομπών οχημάτων. Από το 2000 λοιπόν έχουμε αποκομίσει μια σημαντική εμπειρία του κοινού κέντρου ερευνών για τα θέματα αυτά και έχουμε φτάσει τώρα ένα επίπεδο τεχνολογικής αριστεία που είναι γενικά αναγνωρισμένο από, από όλους. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα των εκπομπών. Μας έχουν ζητήσει και έχουμε αναπτύξει και δικές μας πρωτοβουλίες για τον για την έρευνα των εκπομπών και των μικροσωματιδίων και από αυτή την άποψη ξεκινήσαμε το έργο μας πολύ σύντομα από την, μετά από τη δημιουργία του εργαστηρίου για τα βαρέα οχήματα και επί τη βάση αυτής της γνώσης που συλλέξαμε συνεχίζουμε και για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Από το 2007 και επέκεινα όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες ε, μετρήσεις εμείς έχουμε πάντα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα το 2007 λοιπόν που έγιναν οι πρώτες μελέτες δημοσιεύτηκαν αμέσως τα στοιχεία αυτά. Όλοι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήξεραν, είχαν τα ίδια δεδομένα που είχαμε και εμείς, τα οποία φάνηκαν και σε δύο μεγάλες εκθέσεις και ήταν σαφές ότι υπήρχε αναντιστοιχεία μεταξύ των εκπομπών στο εργαστήριο και των εκπομπών στο δρόμο, που έδωσαν λαβή και στις τρέχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Είναι φανερό λοιπόν, ήταν ήδη φανερό ότι υπήρχε κάποιο συστημικό πρόβλημα στις μετρήσεις εργαστηρίου. Εστιάζαμε λοιπόν σε αυτό και εδώ πρέπει να το δούμε σε από κάποια απόσταση. Όλη η εμπειρία μας στο κοινό κέντρο ερευνών βασίζεται μονάχα σε 20-25 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ζόρτζο. Από τα άτομα αυτά λοιπόν είναι κεφαλής μονάδος. Αυτή η μικρή μονάδα θα έπρεπε να εστιάσει στην προτεραιότητα που ήταν μια συστημική προσέγγιση και η εξέβρεση μιας συστημικής λύσης. Επομένως, να βρούμε μια νέα μεθοδολογία που να αντικαταστήσει την προηγούμενη μεθοδολογία που δεν λειτουργούσε σωστά και να προχωρήσουμε προς τη μέτρηση πραγματικών εκπομπών σε κανονικές συνθήκες οδήγησης. Αυτό βέβαια δεν ήταν δεδομένο πριν από 2-3 χρόνια. Χρειάστηκε να αγωνιστούμε για να πιέσουμε, να πείσουμε ότι η μέτρηση των εκπομπών στον δρόμο είναι η πραγματική λύση για το πρόβλημα αυτό και τελικά αυτό επελέγει ως και η λύση και θα περάσει στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα αυτοκίνητα οχήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έρχομαι τώρα στη τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Όπως ξέρετε υπήρξε το σκάνδαλο με την Volkswagen στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε αυτή η αποκάλυψη και η παραδοχή από την πλευρά της Volkswagen έναντι της EPA, της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι υπάρχει αναντιστοιχεία μεταξύ της λειτουργίας των συσκευών στο εργαστήριο και στον δρόμο. Εδώ έχουμε λοιπόν το δεύτερο κομβικό σημείο, τη δεύτερη μεγάλη ε, στιγμή που βλέπουμε να δημιουργείται, να έρχεται ανάγλυφο το πρόβλημα αυτό και η Κομισιόν ε, προσπάθησε να το αντιμετωπίσει αυτό με την πρότασή της που διατύπωσε τον Ιανουάριο του 2016. Οπότε με την πρόταση αυτή γίνεται σαφές ότι η ανεξάρτητη επαλήθευση της έγκρισης τύπου και έλεγχη σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα πρέπει να είναι ο δρόμος με τον οποίο θα ακολουθήσουμε. Και από τότε εμείς εργαζόμαστε για να δώσουμε την απαραίτητη υποστήριξη για την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήν ώστε να καταλήξουμε στην κατάλληλη νομοθεσία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανέλαβε και αυτό το πρόσθετο καθήκον της ανεξάρτητης επαλήθευσης και εξασφάλισης της διαφάνειας των διαδικασιών έγκρισης τύπου. Αυτό τώρα λοιπόν είναι και κομμάτι της νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν και ελπίζουμε ότι σε ένα χρόνο θα είμαστε σε θέση ήδη να κάνουμε τις απαραίτητες δοκιμασίες για τις συσκευέ μέτρησης. Έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη, μπορούμε <clears throat> να ξεκινήσουμε ήδη αύριο μια πρώτη φάση να ελέγχουμε 30-40 αυτοκίνητα και σε δύο χρόνια μπορεί να φτάσουμε σε 100-130 οχήματα το χρόνο. Το κόστος σε επίπεδο προϋπολογισμού θα είναι περιορισμένο, περίπου 9 εκατομμύρια και έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε αυτά τα οποία κάνει η EPA στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τον αριθμό των οχημάτων που ελέγχονται και πιστεύω ότι και η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να δράσει εάν παρατηρηθεί μια, μια διαφορά, μια απόκληση μεταξύ των τιμών που μετρούνται. Επομένως το μήνυμά μου είναι ότι έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτό το είδος εργασίας Σα είπα για του ε, γενικά προτροποποιημένου οργανισμού, σαν παράδειγμα. Μια περίπτωση που αν έχουμε μια εντολή από την Κομισιόν είμαστε πάντα έτοιμοι να δράσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Κάνουμε τέτοιο έργο με την ε, έκθεση τη Κομισιόν και όταν υπάρχει η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Θα χρειαστούν δύο χρόνια μονάχα για να μπορούμε να λειτουργούμε με ε, την πλήρη ικανότητά μας. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν κυρία Πρόεδρε, θα είμαι έτοιμος να απαντήσω και επίσης και ο συνάδελφος μου Τζοβάνι Τισάντη είναι εδώ αν ε, υπάρχουν τεχνικά ερωτήματα. Έχω και τον Γιώργιο Μαρτίνη, ο οποίος είναι ο αρχηγός μονάδος για τα οχήματα και μπορεί και αυτός να με βοηθήσει. Περνάμε τώρα στην ακρόαση. Καταρχήν ο εισηγητής, ο κύριος Γκίζεκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας που ήρθατε σήμερα εδώ. Είχαμε και μια πολύ καλή επίσκεψη στην Ίσπρα που απαντήσατε σε ερωτήσεις και είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε την αλληλογραφία του Κοινού Κέντρου Ερευνών με την Κομισιόν. Εν τω μεταξύ έχουμε την αλληλογραφία. Έχω εδώ απόσπασμα της 17ης Δεκάτου 2000 16 όπου αναφέρεται ένα email του Απριλίου 2012 που αφορά το ζήτημα των εκπομπών οξυδίου του αζότου μεταξύ 20 και 30 βαθμών. όπου είναι χαμηλότερες οι εκπομπές. Και εκεί πέρα η αρχή σας μιλάει για το λεγόμενο cycle beating και ένα memory effect. Η απάντηση της Κομισιόν στο email σας κάνει λόγο για hard cycle beating. Το ε, cycle beating δεν είναι ούτως ή άλλως νόμιμο. Ε, ή μάλλον δεν έχει οριστεί ε, νομικά, με συγχωρείτε. Δεν είχατε την υποψία πως, έχετε, πως βρίσκεστε απέναντι σε μια παράνομη διάταξη που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 Οπότε το email πρέπει να αντιληφθείτε ότι κάθε μήνα έχουμε 2 εκατομμύρια email. Με την υπόλοιπη κομισιόν. Για το συγκεκριμένο ε, που λέτε ότι το cycle beating δεν είναι ένας καθαρνομικά καθορισμένος όρος. Αφορά πράγματι βελτιστοποίηση του κύκλου και αφορά διάφορα ζητήματα. Αλλά στο συγκεκριμένο αυτό όχημα δεν μιλάμε για το όχημα το οποίο ε, είναι στην αγορά. Μιλάμε για ένα πρωτότυπο το οποίο αφορούσε τις ε, μετρήσεις διοξιδίου του άνθρακα. Και το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι τα ευρήματα αυτά δεν εμφανίστηκαν το 2016. Αυτό ήταν ε, νομίζω τρεις μέρες μετά τα ευρήματα, αν δεν κάνω λάθος, ε, μετά από το email αυτό, παρουσιάστηκε το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή και επίσης τα δεδομένα αυτά υπάρχουν στην έκθεση, οπότε δεν είχε κρυφτεί κάτι, αλλά είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Για τα υπόλοιπα οχήματα που είχαν αναλυθεί, ε, ήταν τα οχήματα τα οποία πήραμε από, την εταιρεία, από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν ε, πρωτότυπο. Ήταν στην φάση των δοκιμών ακόμα. Να είναι σαφές είναι ένα πρωτότυπο. Παρόλα αυτά βρήκατε πως υπήρξε αυτή η βελτίωση στα οξύδια του αζότου και αναρωτιέμαι όταν διαβάζει κανείς για cycle beating και hard cycle beating ε, γίνεται περίεργος. Εσείς να αναρωτηθήκατε πως υπάρχει κάποια παρανομία όταν έχουμε τέτοια περίεργα αποτελέσματα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε και την συζήτηση εδώ πέρα για τη νέα οργάνωση της ε, έγκρισης τύπου και της εποπτείας της αγοράς. Συζητάμε για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, για ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών. Ποιος είναι ο δικός σας ο ρόλος. Θεωρείτε ότι το GRC θα είναι μια αποκεντρωμένη υπηρεσία, μια υπεραρχή στην Ίσπρα θεωρείται ότι πρέπει να οργανωθούν τα πράγματα αποτελεσματικά. Νομίζω είναι σαφές πως δεν θα είμαστε μια υπηρεσία, αλλά θα έχουμε μια δυνατότητα υποπτίας όπως έχουμε και σε άλλους ε, κλάδους, ίσως να ενισχυθεί κάπως εδώ. Οπότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε αυτά τα πράγματα και η Κομισιόν θα έχει τις αρμοδιότητες να ρωτήσει ε, ότι το αμάξι αυτό, ξέρω εγώ, συμπεριφέρεται περίεργα. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν πολλές ε, στρατηγικές ε, για να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση. Αν υπάρχει διαφάνεια και νόμιμη πρόσβαση στα έγγραφα του κατασκευαστή, ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει γιατί υπάρχει μια περίεργη συμπεριφορά. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ω δυνατότητα. Και χωρί την συνεργασία των κατασκευαστών χωρίς όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για αυτό το σκοπό. Δεν μπορούμε να ερευνήσουμε. Νομίζω λοιπόν πως θα έχουμε σοβαρές αλλαγές στο, στο μέλλον με την ε, δυνατότητα αυτή. Ο κύριος Χερμπράντη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας ε, κύριε Σούτσα. Θα ήθελα να επανέλθω στην ακρόαση που είχαμε πριν από λίγους μήνες με την κυρία Αντελιάηλα Αλκουντέρη. Και ένα ζήτημα το οποίο δεν επιλύθηκε είναι ότι το Κοινό Κέντρο έρευνων βρήκε στις μελέτες κάποια περίεργη συμπεριφορά κάποιων αυτοκινήτων και δεν έγινε κάποια άλλη μελέτη μετά. Η απάντηση ήταν ότι δεν μας ε, έδωσε η Γενική Διεύθυνση χύψει την εντολή. εγώ έμαθα ότι η αρχική έρευνα με την οποία τα βρήκατε ήταν μια μελέτη ιδίας πρωτοβουλία, όπως λέμε. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Τι εννοείτε. Οι επόμενε μελέτε υπήρχαν δύο ε, μελέτες και η συνέχεια αποδόθηκε ήταν σαφή στο πλαίσιο της ε, ρυθμιστικής ε, διαδικασίας. Η μελέτη στην οποία υπενηχθήκατε πράγματα τα οποία πήγαιναν πέρα από τον ξεπεράσει κανείς τον κύκλο δοκιμών και μιλούσατε για διατάξεις ε, αναστολής. Και νομίζω πως οι επιστήμονες συνεχίζουν να ερευνούν μέχρι να καταλάβουν το τι συμβαίνει. Αλλά το JRC μάλλον δεν το έκανε και μας είπατε ότι δεν, σε έδωσε εντολή η Κομισιόν, αλλά η μελέτη η οποία βρήκε αυτές τις αποκλήσεις, εμένα μου είπαν ότι ήταν δική σας πρωτοβουλία και ότι μπορείτε να κάνετε μελέτες, έρευνες, χωρίς να σας το έχει ζητήσει κάποια γενική διεύθυνση. Το ερώτημά μου είναι, ισχύει κάτι τέτοιο και αν ναι, γιατί δεν αναλάβετε και άλλες πρωτοβουλίες να δείτε το ζήτημα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε, ναι, το κάνουμε αυτό ε, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλία και οι συνάδελφοί σας έχουν τη δυνατότητα ε, να το δουν, ε, όπως παραδείγματο χάρη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί σε 10 χρόνια θα έχουμε την ίδια κατάσταση με τώρα. Για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οπότε το κάνουμε αυτό προφανώς, αλλά εδώ δεν είναι μια εντολή, αυτή είναι η παρεξήγηση μάλλον, δεν μιλάμε για εντολή προς το κοινό κέντρο ερευνών, μιλάμε για εντολή προς την Κομισιόν, όπως εξήγησα στην εισαγωγή μου, ίσως δεν ήταν σαφές. Το 2014 που πήγα εγώ, μέχρι Εκ τότε δεν νομίζω να υπήρχε κάπου η υπόνοια ότι υπήρχε αυτή η διάταξη αναστολής. Θα σας διαβάσω από μέσα. Έχουμε την περίληψη από τον Νοέμβριο του 2015, χρόνια πριν το σκάνδαλο 2010. Αυτό είναι δικό σας. Όμως ένα όχημα το οποίο δοκιμάστηκε έδειξε εξαιρετικά υψηλέ ε, εκπομπές οξυδίων του αζότου στο δοκιμές τύπου 6. Εφόσον οι δοκιμές ε, τύπου 6 αυτή τη, ρυθμή, τη στιγμή δεν ρυθμίζονται, έχουμε εδώ πέρα μια υπόνοια πολλής πολύ περίεργης στρατηγικής για να ξεπεραστεί ο κύκλος, ε, για να παρακαμφθεί ο κύκλος. Ερωτηματικό. Δηλαδή, ήδη από τον Νοέμβριο του 2010 ήταν σαφές για εσάς ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, ότι υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά οχημάτων που πήγαινε πέρα από την κανονική ας πούμε, προσπάθεια να περάσει ένα μάξιο κύκλο δοκιμών όταν, έχετε, όταν είχατε κάτι παραπάνω από μια υπόνοια ή αίσθηση, είχατε σχεδόν αποδείξεις παρανομίας. Όχι αν είχαμε αποδείξεις ε, παρανομίας, προφανώς θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Γιατί, εξ όσων γνωρίζω, μια στρατηγική διάταξη δεν είναι παράνομη. Μια διάταξη αναστολής είναι παράνομη εγώ σας διαβάζω από μέσα, από την περίληψη των ευρημάτων. Τέλος πάντων, δεν θέλετε να απαντήσετε. Ε, για την αλληλογραφία ρώτησε ο συνάδελφος και μίλησε για τον Νοέμβριο του 2012. Στο ίδιο email η απάντηση ήταν ε, είναι δυνατόν να περιληφθούν αυτά τα αποτελέσματα στην παρουσίασή σας για την 5η, 30 Μαΐου 2012. Μιλούσατε για κάποια ομάδα εργασία όπου παρουσιάστηκε αυτό. Μπορείτε να μου πείτε πιο λεπτομερό πού παρουσιάστηκε αυτό, σε ποια ομάδα εργασία. Η παρουσίαση έγινε σε μία συνεδριάση της ομάδας για τις μετρήσεις υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης και μετά αναπτύξαμε τη διαδικασία. Ναι, λέγει ο Σχέπνερ, όλοι όσοι είναι εδώ όμω ενημερώθηκαν για τα ευρήματα. Ο κύριος Κάρνης έχει το λόγο. Ευχαριστούμε όσο προχωράμε τόσο βρίσκουμε. Πότε το Κοινό Κέντρο Ερευνών συνειδητοποίησε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ε, εργαστηριακών από τη μία και από την άλλη των ε, πραγματικών δοκιμών όσον αφορά το διεξίδιο του αζόντου. Όταν αρχίσαμε τις δοκιμές, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές. 2007. Το 2007 αρχίσατε να επισημαίνετε αυτές τι διαφορέ με προσεκτικά το διαπίστωσε ο συνάδελφος αν ήταν κάτι το παράνομο. Εγώ εδώ θα σταθώ σε αυτές τις διαφορές. Το 2007 ε, είναι μακριά λίγο, μας τον όλοι πιο νέοι, υγιέστεροι και τα πνευμόνια μας καλύτερα. Και τι έγινε. Ε, ανήκυψαν κάποια ζητήματα, χτύπησε κανένα καμπανάκι. Τι κάνατε. Το 7 είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα. Όπως ξέρετε, για το RDE είχαμε τότε πολύ καινούργια την τεχνολογία, για τα επιβατικά, οπότε και έπρεπε να γίνει περισσότερη ανάλυση. Ακριβώς αυτό μας απασχόλησε σε αυτή την ανάλυση και έτσι καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα το 2010. υπήρξε ένα κατάλογο των ε, αυτοκινήτων που δοκιμάστηκαν και ξαναδοκιμάστηκαν. Πολύ σημαντική στιγμή αυτή, τον Ιούνιο του 9, που είχαμε τα αυτοκίνητα προδιαγραφής Euro 5. Οπότε αφού τα καινούργια αυτοκίνητα είχαν την ίδια συμπεριφορά, θα πρέπει να δούμε αν ισχύει αυτό ή αν υπήρξε βελτίωση. Υπήρξε βελτίωση του κ. Κάριν. Όχι, απάντησε. Άρα από το 7 μέχρι το 9 και το 10 εξετάζεται τα πράγματα, μία μελέτη μετά την άλλη και ότι ακόμα υπήρχαν κάποιε διαφορέ, οπότε ακόμα ναι, το 10, τι κάνατε. Το 10 είχαμε αυτό το διάσημο εργαστήριο στο οποίο τον Νοέμβριο. Προσφέρθηκαν όλα τα αποτελέσματα και έλαβε απόφαση η Κομισιόν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει πρόβλημα συστημικό για την μεθοδολογία των δοκιμών η οποία είπαν πρέπει να αντικατασταθεί το δε Ιανουάριο του 11 συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα εργασία και όπως σας είπα δεν ήταν τότε και τόσο σαφές ότι η μεθοδολογία που εμείς προτείναμε επρόκειτο να γίνει αποδεκτή από όλους. Τότε υπήρχαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Και εμείς είχαμε διαλέξει σαφώς πιο προτιμούσαμε. Και τέλος, το 14 πέρασε αυτό το σενάριο, αλλά όχι το 11. Γιατί ακριβώς υπήρχαν διχογνωμίες ακόμα και μεταξύ των επιστημόνων. έλεγε, άλλοι θέλανε το modeling, άλλοι θέλανε το αμερικάνικο πρότυπο. Τέλο πάντων, ε, υπήρχαν πολλή, έγινε πολύ κουβέντα για αρκετό καιρό, μέχρι ότου να πιστεί ο κόσμο για το ποια είναι η σωστή προσέξη. Κάριν, καλώ. Το 7 λοιπόν ότι κάτι. Γίνεται το 10 ε, φτιάξατε αυτό το εργαστήριο και το 14 τελικά υιοθετήθηκε το σενάριο που θέλατε Ίσως τότε κάτι αλλάξει. Το 17, α, μια δεκαετία και ούτε. Όταν δημοσιοποιήσατε τις μελέτες, δεν αναρωτήθηκε κανένας γιατί αφού αυτά γίνονται στο ντίζελ, γιατί να μην γίνονται τα ίδια και στους βενζινοκινητήρες. Ο άλλος κύριος. Ναι, γνωρίζαμε τότε ότι οι ντίζελοκινητήρες έχουν ένα σύστημα πολύ αποδοτικό για πάσα συνθήκη λειτουργίας. Αν δεν ανατρέξετε στο παρελθόν, θα δείτε ότι είχαμε διαφορετικά πρότυπα για τους διζελοκινητήρες. Και ήδη ο νομοθέτης για το γύρο 3 και 4 είχε συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται χρόνος ούτως ώστε για όλα τα οχήματα να υπάρχουν κάποια συστήματα after treatment. Ναι, Κάρινς, όμως ε, τα πνευμόνια μας ε, αρρώστηναν, αλλά δεν αρωτήκατε τότε γιατί να μην εξελίξετε τους κινητήρες, τους διζελοκινητήρες, κάτι να γίνει. Ναι, τα πρότυπα επέτρεπαν για τους διζελοκινητήρες ε, χειρότερες εκπομπές. Κύριε Ντάνης. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να καταλάβω αυτό το τελευταίο σημείο που είπατε, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε γιατί δεν υπήρξε ποτέ ανησυχία για τα θέματα αυτά, επειδή δεν έχετε κάποια εντολή από την Κομισιόν να ερευνήσετε ή γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία ότι υπήρχαν συσκευέ αναστολής, διατάξεις αναστολής η κυρία Αλ Χαουνταρή είπε ότι δεν υπήρχαν ανησυχίες γιατί δεν υπήρχαν ε, στοιχεία. Και είπατε εσείς ότι δεν υπήρχε εντολή. Ποιο από τα δύο ευσταθεί. Δεν είχαμε στοιχεία που να δείχνουν ότι υπήρχαν διατάξεις αναστολής. Γιατί για να ξέρετε αν υπάρχουν διατάξεις αναστολής θα πρέπει να έχετε τη συνεργασία του κατασκευαστή ή των αρχών έγκρισης τύπου. Μία συσκευή, μία διάταξη αναστολής είναι λογισμικό, δεν είναι ένα εξάρτημα Και αναφέρθηκε πολλές φορές από πάρα πολλούς ανθρώπους και στην Επιτροπή σας ακόμα, ότι χωρίς την πλήρη συνεργασία των ε, κατασκευαστών δεν μπορεί κανείς να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ναι, λέτε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία. Αν υπήρχαν στοιχεία όμως, θα είχατε κάνει περαιτέρω έρευνες για αυτές τις συντετάξεις αναστολής. Χρειάζεστε την τεχνολογία, <clears throat> μια μεθοδολογία για να μπορείτε να ελέγξετε αν οι υποψίες σας ευσταθούν. Αν έχετε μια συμπεριφορά η οποία δεν οφείλεται στον κύκλο δοκιμασίας, μπορεί να έχει κανείς υποψία, αλλά δεν έχει μια απόδειξη. Μα αυτό όμως θα έπρεπε να οδηγήσει σε περισσότερα ερωτήματα. Αν είχατε μια μεθοδολογία ανεπτυγμένη τότε, τότε θα μπορούσατε να προχωρήσετε σε αυτό. Αλλά εκεί είναι η εντολή της ε, Κομισιόν. Θα έπρεπε η Κομισιόν να έχει μια εντολή αντίστοιχη με αυτή που είχε η EPA στις ΗΠΑ. Οπότε είναι το, η εντολή ή τα στοιχεία. Γιατί στην αρχή είπατε τα στοιχεία. Ναι, πρέπει να έχετε μια εντολή για να αναπτύξετε τη μεθοδολογία πώς θα ψάξετε να βρείτε δυνητικές διατάξεις αναστολής και μετά μπορείτε να τα ελέγξετε. Μα... Μια στιγμή, λέτε ότι αν είχατε υποψίες ή στοιχεία θα είχατε κάνει περαιτέρω μελέτες. Μας είπε ο κ. Χερμπράντ για την έκθεση που έγινε τα email της 30 Απριλίου του 2012 και υπήρχαν και περισσότερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010 που αναφέρονται στην παράδοξη συμπεριφορά των οχημάτων. Έχουμε το email της 4 Απριλίου 2008 που εκπεφρασμένα θέτει το θέμα στρατηγικών αναστολής και διατάξεων αναστολής και κάπου λέγεται αυτή ακριβώς η έκφραση «Defeat strategy ή device μέσα σε αγγείλες στο κείμενο. Γιατί όλα αυτά δεν ήταν επαρκή για να προχωρήσετε σε περαιτέρω έρευνες βάσει της εντολής σας ω κοινό κέντρο έρευνων. Νομίζω ότι υπάρχει κάθε λόγος να προχωρήσετε σε περαιτέρω έρευνες. Αυτά όλα ήταν σε γνώση των μελών του κοινού κέντρου ερευνού, ερευνών και γιατί εσείς δεν δώσατε συνέχεια. Μα είναι σαφές λέει ο κύριο Σούσα από τις μελέτες μας ότι υπάρχει ένας κατάλογος οχημάτων diesel που δείχνουν αναντιστοιχίε μεταξύ πραγματικών συνθήκων και κύκλου δοκιμών. Είναι πολύ λοιπόν λογική η... το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα. Οι συσκευές αναστολής δεν είναι συστημικό πρόβλημα. Ή αλλιώς μπορείτε να πείτε ότι όλοι οι κατασκευαστές κοροϊδεύουν τον, ε, την έγκριση τύπου. Ναι, αλλά Εάν εσείς έχετε την υποψία ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν θα έπρεπε εσείς να κάνετε κάποια έρευνα και να καταλήξετε σε συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι συσκευή διάταξη αναστολής γιατί α, β και γ. Ναι, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ακόμα και η οι στις πολιτείες δεν μπόρεσε να εντοπίσει κάποιες συσκευές, κάποιες διατάξεις αναστολής μέχρι να τους το πει η Volkswagen. Ναι, αλλά αυτό το ανακάλυψε η Volkswagen διότι είχε περίεργεια η EPA και του ανάγκασε να αποκαλύψουν την πραγματικότητα. Αλλά γιατί δεν είχε το κοινό κέντρο έρευνα την αντίστοιχη περιέργεια. Εμεί ζητήσαμε από την Κομισιόν μια τέτοια εντολή τον Ιανουάριο, αλλά δεν έχουμε ακόμα την εντολή να κάνουμε αυτό που κάνει η EPA στι ΗΠΑ. Θα ήταν δύσκολο. Οπότε λέτε πάλι ότι πρόκειται για την εντολή. Λοιπόν, είναι πολύ μπερδευτικά αυτά που λέτε. Πότε λέτε τα στοιχεία, πότε είναι η εντολή αν θέλει κανείς να ερευνήσει για, για διατάξεις αναστολής, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβετε τι γίνεται, τι έγινε το 2010 με τη γνώση που έχουμε το 2016. Αν δείτε πόσα διαφορετικά οχήματα έχουν ελεγχθεί, βλέπετε ότι υπάρχουν αναδυστυχίες και θα ακολουθήσετε την πιο ορθολογική άποψη λέγοντας ότι δεν στέκει η μεθοδολογία να ακολουθήσουμε μια άλλη μεθοδολογία. Χρειάζεται μια συστημική λύση. Τι θα κερδίζαμε ακόμα και αν αποδεικνύαμε ότι υπάρχουν, υπάρχουν αυτοκίνητα με, με διατάξεις αναστολής. Απλώς βλέπετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο. Να χρησιμοποιώ το χρόνο μου και το ξεπέρναω. Ακόμα είμαι μπερδεμένος είναι η εντολή, είναι η έλλειψη στοιχείων. Ποιος είναι ο βασικός παράγων πίσω από την έλλειψη ικανότητά σας να συνεχίσετε τις μελέτες σας. Καταλαβαίνω τι δυσκολίες που μας αναφέρατε και σε έχετε αναφέρει. Είναι και τα δύο και η εντολή και τα στοιχεία. Δεν είχατε ούτε στοιχεία ούτε εντολή. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι ξέρατε τότε. Ναι, θέλω να σας πω ότι δεν είχαμε στοιχεία και δεν είχαμε κανένα λόγο να κάνουμε έρευνα για, για διατάξεις αναστολής, γιατί δεν είχαμε κάτι το οποίο να υποδεικνύει την ύπαρξη διατάξεων αναστολής. Γι' αυτό εμείς προχωρήσαμε προς μια συστημική λύση. Και αν απαντώ το υποθετικό σας ερώτημα, ακόμα και αν είχαμε την υποψία ότι υπήρχαν διατάξεις αναστολής, δεν θα μπορούσαμε να πάμε να τα ψάξουμε αυτά, γιατί δεν θα είχαμε την εντολή δεν θα είχαμε την πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα των κατασκευαστών ή των αρχών έγκρισης τύπου. Είναι υποθετικό αυτό ε, ερώτημα το οποίο απαντώ. Εμείς θέλησαμε να δώσουμε μια συστημική λύση η οποία θα ξεπερνούσε το θέμα των διατάξεων αναστολής γιατί για μας με 20 άτομα ήταν σημαντικό. Υπήρχαν ερευνητέ σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλά είχαν δημοσιευθεί μέχρι το 2007. Γιατί δεν είχε βρει κανεί τι διατάξει αναστολή αν ήταν τόσο απλό. Τούρμε. Διαδικαστικό. Μπορούμε να κάνουμε, να τραγουδήσουμε για 30 δευτερόλεπτα το Happy Birthday για το Step Dance. Η κυρία Μάσινα. Ευχαριστώ. Στα γερμανικά. Βάλτε τα ακουστικά σας λοιπόν. Όπως είπατε προηγουμένως, η εντολή σας είναι να υποστηρίζετε την Κομισιόν επιστημονικά για το έργο της. Πολύ καλό είναι αυτό να έχει αυτή την υποστήριξη η Κομισιόν. Αλλά για μας είναι πάντα αυτό το ερώτημα. Η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Αν το 2007 υπήρχαν κάποια προβλήματα που είχατε δει με τις εκπομπές οξυδιών του άζωτο και είχατε ήδη το 2010 σαφείς ενδείξεις στο εργαστήριο που έγινε, μήπως θα έπρεπε να το φέρετε σε γνώση της Κομισιόν, να ξέρει όλα αυτά τα πράγματα η Κομισιόν. Και αν έγινε αυτό το πράγμα, ποια ήταν η αντίδραση της Κομισιόν, πώς αντέδρασαν και τα κράτη-μέλη στις ειδήσει αυτές που θα μπορούσαν να τους είχατε δώσει, ότι πράγματι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την εφαρμογή της νομοθεσίας ήδη το 2007. Όλα αυτά τα βρήματα, όπως σωστά είπατε, παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο. Οπότε δύο μήνες μετά φτιάξουμε την ε, ομάδα εργασίας για ακριβώς για αυτό το πρόβλημα. Οπότε έτσι έχουμε το καινούργιο οργανιστικό πλαίσιο για τις RDE. Ε, Επομένως, ήμασταν πρωτοπόροι παγκοσμίω. Διαλέξαμε δηλαδή να γίνει νόμος ε, αυτού του είδους η μέθοδος. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά η Κομισιόν. Όχι, όχι. Δεν σα ρώτησε αν τα πήγατε καλά ω Κομισιόν. Εσείς είστε ο φύλακας των συνθήκων. Το 10 έγινε αυτή η ενημέρωση και οι επιστήμονες το ήξεραν έτσι και δεν έγινε όμως τίποτα. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Να μια διαφοροποίηση μεταξύ defeat device και defeat strategy. Το 10 είχατε δει μια στρατηγική σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, αυτή η διάταξη. Τι έκανε η Κομισιόν για να αλλάξει κάτι. Κάνατε κάτι. Απάντησε. Ας ε, επιστρέψουμε σε αυτόν τον περίφημο ορισμό για τη στρατηγική τη συνάντηση του Νοεμβρίου του 10. Τότε αναφερθήκαμε στα τεστ σε πλην 7 βαθμούς ακριβώς όπως προέβλεπε ο νόμος. Όμως δεν ζητούσε στους μειών 7 να μετρηθεί το οξύδιο του αζόντου. Δεν προβλεπόταν κανέ, καμία ωριακή τιμή για το νόξ στους πλήν βαθμούς και διαπιστώθηκε ότι κάποιο αυτοκίνητο σε αντίθεση με άλλους διζελοκινητήρες κάποιο αυτοκίνητο παρουσίασε μια διαφορά μεταξύ εκπομπών στη μέτρηση των 20-25 βαθμών σε σχέση με τον όξ, σε σχέση με την μέτρηση στους πλήν 7 βαθμούς. Οπότε έτσι καλύπταμε την οριακή τιμή που αφορούσε ορισμένες μόνο εκπομπές. και υπήρχε μεγαλύτερη εκπομπή στο ξεκίνημα με κρύο τον κινητήρα. Οπότε γι' αυτό και δεν δημιουργήθηκε καμία υποψία σε σχέση με τη διάταξη αναστολή. Υπήρχε βέβαια αυτή η ένδειξη ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει για τον όξ του πλήν 7. Άλλη ερώτηση. Μα είπατε ότι η διάταξη αναστολής δεν επισημάθηκε από την EPA. Είναι δυνατόν να, να τους εντοπίσουν οι επιστήμονες. Όχι, δεν το κάναμε ποτέ αυτό, ο κύριο Σούγα. Αλλά τώρα αναπτύσσουμε μία μεθοδολογία που μας δώσει τη δυνατότητα να επισημάνουμε ύποπτα οχήματα. Να τα εντοπίσουμε. Τώρα, όσον αφορά την νομοθεσία, σήμερα αν υπάρχει κάτι το ύποπτο, η μόνη αρμόδια αρχή είναι η αρχή έγκριση τύπου του κράτου μέλου. Και να πάει στην αυτοκινητομηχανία για να πει γιατί χρησιμοποίησε αυτή τη στρατηγική για την προστασία τη μηχανή. Μπορείτε να το δικαιολογήσετε, μπορείτε να μας παράσχετε τα τεχνικά στοιχεία γιατί το διαλέξατε και πώς λειτουργεί. Οπότε τότε εκείνη η αρχή μπορεί να κρίνει κατά πόσο είναι διάταξη αναστολής ή κατά πόσο είναι μια στρατηγική νόμιμη για προστασία του κινητήρα από τον κατασκευαστή. Αλλά χωρίς τεχνική τεκμηρίωση δεν γίνεται. Εσείς δεν έχετε καμία σχέση με τις εθνικές αρχές. Σχέση μεταξύ και των εθνικών αρχών δεν ενημερώθηκαν για το εργαστήριο. Φυσικά όλοι, όλοι ενημερώθηκαν. Γιατί είπαμε ότι είχαμε τις δημοσίες του 2007, είχαμε κατόπιν αυτή την ε, ε, έκθεση 11-13 που παρουσιάστηκε στο εργαστήριο. Οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν παραστεί. Και η συνέχεια θα μπορούσε να είναι η θέσπιση αντίστοιχη νομοθεσία από την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε, μπορείτε να μας πείτε ακόμη μια φορά. Έχω καταλάβει καλά το τι έγινε. Το 2013 δημοσιεύσατε μια έκθεση που αφορούσε τα προβλήματα μέτρησης ε, της ε, θερμοκρασίας και είπατε στην ε, Κομισιόν ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο χωρίς να κάνετε αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά. Μετά είπατε ότι συνεργάζεστε στενά με την Κομισιόν και μετά στις συζητήσεις αντιληφθήκαμε όλοι ο όσοι δούλεψαν πάνω στο θέμα, στο JRC. Είναι ουδέτεροι και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ε, δεν ε, τίθεται κανένα ζήτημα. Αλλιώς μας παραπλανείτε όλους. Γιατί συνέβη αυτό το 2013 γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε κάτι τέτοιο ε, για να αναθεωρηθεί η διαδικασία και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είστε όντως ε, ουδέτεροι. Τι θέλετε να πείτε, τι δεν δημοσιοποιήθηκε, γιατί όλες οι εκθέσεις ε, και σας έχουμε δώσει έναν κατάλογο το είναι δημόσιες. Τι εννοείται δεν δημοσιεύτηκε το 2013, ποιο πράγμα ακριβώς. Ε, δημοσιεύσα το υλικό, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Τι συνέβη με τις ε, πληροφορίες, γιατί δεν συνέβη τίποτα συγκεκριμένο. μέχρι που τελικά ευνηδιαστήκαμε χάρη στη ΣΥΠΑ. Δεν νομίζω ότι δεν συνέβη τίποτα. Μετά από το εργαστήριο του 2010 υπήρξε μία ομάδα για να εισαχθεί ακριβώς, μία ομάδα εργασίας για να εισαχθεί η νέα μεθοδολογία. Αυτά ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2011 και εφόσον αυτή η ομάδα είχε κάποιες δυσκολίες να αποδεχτεί αυτή την μεθοδολογία ε, από την αρχή. Όπως σας είπα υπήρχαν τέσσερις επιλογές που εξετάστηκαν και μετά μας ζητήθηκε να συνεχίσουμε με τις δοκιμές αυτής της μεθοδολογίας και έτσι καταλήξαμε στη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2013 και μετά κατευθείαν στην έγκριση του πρώτου ρυθμιστικού πακέτου. Νομίζω ότι είναι μια λογική αλληλουχία στοιχείων πρώτα και μετά δράσης. Ε, μα, στις ε, συναντήσεις η διάταξη ήταν σαφές ότι χρησιμοποιούσαν μια διάταξη αναστολής. ή κανείς δεν είχε καταλάβει ότι χρησιμοποιούσαν διατάξεις. ναι, ναι, πράγματι. Κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι χρησιμοποιούσαν διατάξεις αναστολής. Δεν υπήρχαν αποδείξεις. Η όλη συζήτηση για τις ε, παρεκκλήσεις αυτές ε, πήγε στην ομάδα εργασίας μεθοδολογίας αποδείχτηκε ότι η μεθοδολογία ήταν λανθασμένη και υπήρχε συστημικό πρόβλημα, το οποίο συστημικό πρόβλημα αρχίσε να το προσεγγίζει η ομάδα και κατέληξε στα πακέτα αυτά της σχετικής ε, νομοθεσίας που στόχο είχε ακριβώς να βελτιώσει την ε, κατάσταση. Γι' αυτό λέω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος ε, παγκοσμίω με αυτή την προσέγγιση. Και τώρα οι άλλοι ακολουθούν το παράδειγμά μας. Κύριος Τούρμας. Μια στιγμή, μια στιγμή. Ε, σύντομα επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ο κύριος ε, Σούκα απάντησε ότι στις 4 Μαΐου υπήρξε και ένα email ε, στην ομάδα εργασίας ε, σύμφωνα με τα όσα μας είπε η Κομισιόν υπήρχε μόνο μία ομάδα εργασία στις 24 οπότε στις, 12, στις 3 Μαΐου 2012 υπήρξε και άλλη μία ομάδα εργασίας τι συνεδρίαση ήταν αυτή αν μπορεί να μας εξηγήσει ο κ. Σούκα Συγγνώμη, δεν θυμάμαι όλα τα στοιχεία, όλες τις λεπτομέρειες της ε, συνάντησης θα τα ελέγξουμε και θα σας τα διαβιβάσουμε. Ελέγξτε τα και πέστε μας, λέει η Ευχαριστώ κύριε Σούτσα. Στην απάντησή σας, λέει ο κύριος Τούρμες, στο ερώτημα υπαριθμών 8, λέτε ότι η δημοσίευση της επίσημης έκθεσης οδήγησε σε μια διαδικασία αναθεώρησης. Υπάρχουν κάποια, υπάρχει κάποια ανταλλαγή email σε αυτή την εσωτερική διαδικασία αναθεώρησης μεταξύ της DG Enterprise και, της, του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Πώς γίνεται, υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν emails. Στείλατε αυτή την έκθεση στην ε, DG Enterprise, σας απέστειλε κάποια email από εκεί, η DG Enterprise ή όχι. Όλα τα emails τα οποία έχουν να κάνουν αυτό το θέμα σας έχουν δοθεί. Είναι 300, 300 έγγραφα συνολικά. Δεν ξέρω ποια email ήταν αυτά. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα email για την συζήτηση επί τη βάση της έκθεσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών το 2013. Δεν μπορείτε να μας πείτε ότι κανείς δεν έστειλε ούτε ένα email. Στο σημείο 9, στην ερώτηση 9, λέγατε, από τις δοκιμασίες που γίνανε το 2009, και ο κ. Μαρτίνη ήταν ήδη σε αυτή την ομάδα. Τι είναι λοιπόν από τις αρχές του 2010 μέχρι τον Νοέμβριο. Ούτε ένα email μεταξύ του Κοινού Κέντρου Έρευνων και της DG Enterprise. Πεςτε μου κύριε Μαρτίνη, κανένα δεν στείλατε, ούτε ένα email δεν στείλατε. Μπορείς να, να σας πω, θα πρέπει να ελέγξω με τον συναδελφό μου, ο οποίος ε, συνέτασε την έκθεση αυτή. Αυτό όμω δείχνει δύο πράγματα, λέει ο κ. Έχουμε την έκθεση. Και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιο ε, έγραψε αυτή την έκθεση. Δεύτερον, είσαστε τμήμα τη ομάδο που έκανε τι δοκιμέ. Ποιο ήταν ο ομόλογο σα στην DJ Enterprise, ο κύριο Στάινγκερ ή κάποιο άλλο. Μα δεν ήμουν κομμάτι τη ομάδο ε, δοκιμασία. Εγώ έκανα άλλε μελέτε τότε και δεν μου στείλανε αντίγραφο οποιασδήποτε ανταλλαγή email. Μα τότε κύριε Σούτσα, έχετε μια ομάδα στο Κοινό Κέντρο Ερευνών που κάνει δοκιμασίες. Μετά μοιράζονται τα πορίσματα με την DG Envy, την DG Enterprise και μας λέτε ότι δεν υπάρχει ίχνος ούτε ενός email. Σας ρωτήσαμε να μας στείλετε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες ανταλλαγές email από το Κοινό Κέντρο Ευνών στις διάφορες γενικές διευθύνσεις από το, την αρχή του 2009 ως το τέλος του 2011. Ούτε ένα email δεν έχουμε από τον Ιανουάριο του 2010 ως τον Νοέμβριο του 2010. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Πρέπει να μας δώσετε αυτά τα email που να αποδεικνύει ότι η DG Enterprise δεν ήθελε το κοινό κέντρο ερευνών να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Και λέτε ψέματα. Υπάρχει ένα email από το Σεπτέμβριο του 2010 που κάποιος ζητάει από το κοινό κέντρο ερευνών να μάθει. Γιατί δεν κάνουμε κάποιους, κάποιες δοκιμασίες όπως αυτές που κάναν τότε οι Αμερικανοί και που έγιναν αυτό το καλοκαίρι όταν ξέραμε πια ότι υπάρχουν αυτές οι διατάξεις αναστολής. Ξέρανε λοιπόν, το είχαν ανθιστεί ότι υπήρχαν διατάξεις αναστολής όλοι και η δικιά σας εφήρη κύριε Σούσα είναι να μας δώσετε αυτά τα email. Λέτε ψέματα ότι μας δώσατε όλα τα email. Μα δεν πήρατε ίσως όλα τα email, λέει ο κύριος Σούτσερ. Σας είπα ότι το κοινό κεντρευνών, βγάζει ένα εκατομμύριο email το μήνα. Μα ούτε ένα δεν πήραμε, ούτε ένα για τις ανταλλαγές απόψεων ανάμεσα σε εσά για τις δοκιμές και την DG Enterprise. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Και εσείς είσαστε υπεύθυνου για το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει αυτά τα email. Γιατί δεν μας τα στέλνετε. Και θέλουμε και τα email σε λειτουργικό επίπεδο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι σωστό ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Πρόσθετη πληροφορία. Πήραμε ένα πρόσθετο email σήμερα το πρωί, λέει η Πρόεδρος. Στείλαμε μάλλον ένα mail ακόμα για να ζητήσουμε και πάλι τα email αυτά που αναφέραμε. Μια στιγμή. Είπε η Κομισιόν ότι ψάχνουν ακόμα. Η Κομισιόν έχει μια στρατηγική, η οποία είναι η εξή. Κάνουμε μια ακρόαση. Δεν μας δίνουν τα αντίστοιχα email. Είναι η πέμπτη ακρόαση που δεν έχουμε πάρει τα emails από την Κομισιόν. Έρχονται οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, λένε δεν έχουμε τις πληροφορίες. Και ίσως το βράδυ από τώρα να μας στείλουν κάποια email. Αυτή είναι μια στρατηγική, κυρία Πρόεδρε, που θεωρώ ότι είναι απόλυτα άδικη έναντι μιας επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να κάνει μια έρευνα και ο κύριος Σούτσα έχει ένα κέριο ρόλο σε αυτή τη στρατηγική να μην μας δίνει η Κομισιόν πρόσβαση σε αυτά τα email. Και ελπίζω ότι δεν είμαι ο μόνος βουλευτής που θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία παραπλάνησης έχει τραβήξει ήδη μήνες και ο κύριος Σούτσα έχει ένα κέριο ρόλο με το να μην μας δίνει την πληροφορία αυτή. Δεν είναι φυσιολογικό να μην έχω κύριε Σούτσα ούτε ένα email. Τι θα μου πείτε γι' αυτό. Κύριε Τούρμες, το μοντέλο μας είναι να βασιζόμαστε σε στοιχεία. Θα ήθελα να ξέρω και τα δικά σας στοιχεία μετά από την ανακάλυψη των συσκευών αναστολής. Τώρα όλοι λένε ότι κάποιος τα ήξερε. Αν μου δώσετε κάποια απόδειξη ότι εγώ έδωσα εντολή σε κάποιον να μη σας δώσει τα email, παρακαλώ δώστε μου τα στοιχεία ότι το έκανα εγώ. Δεν έγινε ποτέ. Από την αρχή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πάντα είπα στους, να δώσουν... Σταματήστε τα λέει η πρόεδρος. Αν έχετε στοιχεία ότι εγώ μπλοκάρισα τα email, δώστε μου τα, στοιχεία αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να αρχίσουμε να φωνάζουμε, λέει η πρόεδρος θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να πάρουμε τα στοιχεία και θα αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Τούρμες, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Είχαμε συναντήσει με την Κομισιόν, όπου εξοργιστήκαμε ιδιαίτερα. Εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειες πιο έντονα για να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έλλη. ευχαριστούμε για τα όσα μας καταθέσατε σήμερα με της Επιτροπής μας. Πιστεύω προσωπικά ότι αυτές οι στρατηγικές ακολουθήθηκαν περισσότερο από κάποια κράτη-μέλη με τη βοήθεια της ε, Κομισιόν. Οπότε φυσικά και εσείς έχετε εμπλοκή με τα όσα έγιναν. Οπότε, κατά τη γνώμη σας, το ότι πέρασαν δέκα χρόνια για να υπάρξει κάποια αλλαγή στις δοκιμές δεν είναι κάτι σαν θρησκευτική προσκόλληση και πίστη και όχι ε, εξέβρεση λύσης και βήμα προς το εμπρός. Τώρα βλέπουμε μια αλλαγή. Και πόσα χρόνια, πάρα πολλά θα περάσουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια βελτίωση ε, στην ατμόσφαιρα από το σύνολο των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Μέσης δεν θεωρείται δεν έχετε προβληματιστεί συζητήσει και σε τεχνικό επίπεδο για κάποια άλλα μέτρα. Κάπως να αναξελίξετε το RDE. Κάτι το οποίο θα βρει σύμφωνα και τα κράτη-μέλη. Σούτσα. Υπάρχει η γενική ομοφωνία για το ποια είναι η καλύτερη λύση για τις δοκιμές. Βεβαίως και η τεχνολογία εξελίσσεται και αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε και αυτό και κάναμε όταν κάνατε την αποστολή. Έχουν τα ηλεκτρικά οχήματα, οπότε πια θα υπάρχει θέμα εκπομπών, αλλά θα υπάρχουν άλλα θέματα, θέματα ασφάλειας. Έχουν σχέση με αυτά τα αυτό. με αυτοκίνητα, με τα ηλεκτρικά οχήματα, τα υβριδικά. Υπάρχουν πάρα πολλούς αισθητήρε, εκατοντάδες στα αυτοκίνητα. Και γι' αυτό το περίφημο Internet of Things έχουμε τώρα χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. Μπήκε και στην ε, νομοθεσία. Τι 10 χρόνια είναι πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη και το πώς ε, μικραίνουν όλα τα εξαρτήματα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχεδόν κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί. Οπότε τώρα θα έχουμε μια καλύτερη ανάλυση, ποιοτική ανάλυση στους ε, ελέγχους, στην υποπτήρια της αγοράς, στις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν μπορώ να σας δώσω μία ημερομηνία συγκεκριμένη, αλλά μέσα στην πενταετία θα δείτε ότι θα μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ περισσότερα. 30. Άρα θα γίνει μεγάλη, μεγάλη αλλαγή. Σα ευχαριστώ. Τελευταία με ρώτηση, λέει κυρία Βε. Που έχει σχέση με τα απάντησή σα. Ε, δεν ήρθα στην αρχή τη ομιλία και έχασα κάποια πράγματα. Αλλά τι ρόλο μπορεί να έχει το κοινό κέντρο εργών για αυτή την καινούργια πρόταση που συζητείτε, για την πιστοποίηση των αυτοκινήτων, για την υποπτία της αγοράς. Τι θα μπορούσε να κάνει το κέντρο ερευνών. Και να λύσει αυτά τα προβλήματα υποπτίας της ε, αγοράς εκεί όπου υπάρχουν τέλο πάντων ελλείψεις αδυναμία. Εάν έχουμε την ε, εντολή που δεν την έχουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από 30-40 αυτοκίνητα που θα αναλύσουμε, θα μετρήσουμε τις εκπομπές τους και θα φτάσουμε όμως στα 130 μέσα σε μια διετία. Αλλά τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει σημαντικό ρόλο να διαρματίσει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από όσα σήμερα σε συνεργασία με τις αρχές εγκριστήπου των κρατών μελών. Όμως δεν έχουμε εμείς νομοθετικές, κανονιστικές αρμοδιότητες όλα γίνονται σε εκούσια, θελούσια βάση. Αναπτύξαμε μεθοδολογίες, μας ζήτησαν, μας πρόσφεραν, τέλο πάντων, ε, καινούργιες δυνατότητες με εξειδικευμένο προσωπικό. Άρα είπαμε, όλα αυτά θα αλλάξουν πολύ σύντομα. Και η πραγματική αγορά, η πραγματική δουλειά για την αποκτήρια τη αγορά θα ξεκινήσει και έτσι να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την έγκριση τύπου, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην νομοθεσία. Νομίζω τέλειωσαν οι ερωτήσεις, αλλά θέλω να ξαναγυρίσουμε στα θέματα των ε, email. Οπότε τότε θα τα ξαναπούμε. Αλλά μια που είστε εσείς εδώ και η Κομισιόν, ε, πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα κενό στην ενημέρωση για μια συγκεκριμένη περίοδο. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος, αλλά θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτό το κενό στην ενημέρωση. Θα σας τα πούμε και εγγράφω αλλά μια που είσαστε εδώ, σας λέω ότι θα πρέπει συντόμως αυτό να το κοιτάξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε πάνω Και βεβαίω όταν ε, υπάρξουν τα email, τότε θα σε υποβάλουμε γραφώ κάποιε επιπλέον ερωτήσει. Και πάλι ευχαριστούμε. Περιμένουμε να έρθει ο κύριο Ντεσάντη. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do some έχετε τον λόγο να κάνετε μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι και από μένα. Ε, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω αυτά τα οποία είπα την προηγούμενη φορά όταν είχατε έρθει στην Ίσπρα. Και όπως ξέρετε βρίσκομαι εδώ πέρα ως πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας και Μεταφορών. Οπότε θα ήθελα να συνοψίσω λίγο τη δουλειά που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να πω τα εξής. Η αποστολή του Ινστιτούτου ήταν πάντα να υποστηρίζει από επιστημονική πλευρά την ανάπτυξη της πολιτικής εντός κομισιών. Δηλαδή στηρίζουμε τις γενικές διεθνείς ανάπτυξης, ενέργειας, κλίματος και ειδικά για τις εκπομπές για το γύρο 5 και γύρο 6 για τα αυτοκίνητα, για τα φορτηγά, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Αυτή ήταν η αποστολή μας. Μετά βεβαίως ξεκινήσαμε όπως ξέρετε στον 20ο αιώνα, στα τέλη του 20ου αιώνα γιατί μας είχε τεθεί το ερώτημα αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο υπάρχει στις είπα ανεξάρτητα δεδομένα με βάση τα οποία να αναπτύξουμε την ε, νομοθεσία. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το εργαστήριο οχημάτων και άρχισε η συνεργασία με τους ε, αυτούς οι οποίοι λαμβάναν τις αποφάσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν κοιτώντα την οδηγία ε, Euro 5 που εστίαζε κυρίως στα σωματίδια γιατί τότε τα νανοσωματίδια υποτίθεται ήταν το βασικό πρόβλημα του ντίζελ. Και συνεχίσαμε το 2003, αρχίσαμε να κοιτάμε και τα PEMS για τα φορτηγά. με τα συστήματα έλεγχου των ε, εκπομπών. Και μετά τι έγινε. Το 2005 όταν είχαμε τελειώσει λίγο πολύ την προετοιμασία του Euro 5 η αρμόδια γενική διεύθυνση μας είπε να δούμε τις εκπομπές πραγματικού, ε, πραγματικής διαδρομής και για τα ε, γεωταχή γιατί βεβαίως δεν υπήρχαν στις σχετικές προδιαγραφέ κάποιες διατάξει για την ποιότητα του αέρα καθώ βλέπαμε το θέμα με, τις, ε, με τα οξύδια του αζότου, από το γύρο 2, 3, 4, 5. Οπότε αρχίσαμε από το 0 να αναπτύσσουμε αυτή την τεχνολογία με βάση ακριβώ το φορητό αυτό σύστημα μέτρησης εκπομπών και για τα γεωταχή. Χρειάστηκαν κάποια χρόνια, ξεκινήσαμε το 2007 να αγοράζουμε και να αναπτύσσουμε τις ε, κατάλληλες ε, συσκευέ μέτρηση. Και ξεκινήσαμε τότε με τα αυτοκίνητα με αυτοκίνητα γύρω 3 και γύρω 4 και μετά γύρω 5 μόλις ήταν διαθέσιμα το 2009 περίπου. Οπότε όπως είπε ήδη ο Βλαντιμίρ τελειώσαμε ε, την πειραματική φάση αρχές του 2010, τέλη του 2009. Οπότε 2010 θα ξεκινούσαμε ήδη την ανάλυση και ήμασταν σε επαφή με τους συναδέλφους και οργανωθήκαμε γιατί συνειδητοποίησαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε την επιστημονική κοινότητα, τους ενδιαφερομένους, τα καρατεμέλη και την βιομηχανία για τις ε, ασυνέπειες αυτές που υπήρχαν μεταξύ των εργαστηριακών δοκιμών και των δοκιμών στον δρόμο. Και ξεκίνησε αυτή η ομάδα εργασίας για τις πραγματικές εκπομπές. Ε, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011, μετά χρειάστηκαν δύο χρόνια για να αποφασίσουμε τελικά να ακολουθήσουμε την γραμμή που θέλαμε με βάση το φορητό σύστημα δοκιμών γιατί υπήρχαν και κάποιες διαφωνίες εντός ομάδας εργασίας και τελικά τον Οκτώβριο του 2012 αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία γιατί όλοι συμφώνησαν ότι αυτό ήταν ο μόνος τρόπος να μετρήσουμε τις εκπομπές στο δρόμο. Αλλιώς θα έπρεπε να ξαναπάμε στο εργαστήριο και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι, είναι πάλι εργαστήριο. Και μετά τον Οκτώβριο το 2012 χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια για να φτάσουμε στην στο πρώτο σχέδιο πρότασης γιατί έπρεπε να αποφασίσουμε τι μεθοδολογία θα χρησιμοποιούσαμε για την αξιολόγηση των δεδομένων και τις συνθήκες της δοκιμής. Οπότε όταν αποφασίζει κανείς να κάνει κάτι πριν φτάσει στην απαραίτητη συνένεση για να περάσουμε στην ε, έγκριση. Χρειάζεται χρόνος να πείσουμε τους ειδικού ε, για να καταλήξουμε σε μια συνένεση. Αυτά χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να φτάσουμε στο πρώτο αυτό πακέτο, το οποίο ψηφίστηκε το Μάιο 2015. Έτσι λίγο πολύ έχουν τα πράγματα το πώς ε, καταλήξαμε εκεί. Και μετά από αυτό, τι κάναμε. Συνεχίσαμε να εργαζόμαστε σε συνεργασία με τους διάφορους ε, ενδιαφερόμενους και φτάσαμε στο επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα. Και μπορώ να σας πω σύντομα τα εξής. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή ε, έχουμε αναπτύξει και είμαστε περήφανοι, να σας πω την αλήθεια, την καλύτερη δυνατή μεθοδολογία για την μέτρηση των πραγματικών εκπομπών και αυτό επαληθεύεται γιατί τώρα αυτή τη στιγμή η Κορέα, η Κίνα αποφάσισαν να εθετήσουν την ίδια μεθοδολογία, οπότε θεωρώ ότι λάβαμε την σωστή απόφαση, να μην χάσουμε πάλι χρόνο, να ψάχνουμε διάφορα τεστ, γιατί ό,τι και να αποφασίσουμε είναι δυναμικές δοκιμές και να κάνουμε κάτι το οποίο είναι επαναστατικό, ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός και στο μέλλον ό,τι και να λέμε, ε, η υιοθέτηση, με την υιοθέτηση τώρα του τεστ πραγματικών συνθήκων θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε να μην σεφαστεί τις προδιαγραφές εκπομπών. Οπότε για εμένα το τεστ αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική θετική απόφαση που στις Κομισιόν και τα κράτη-μέλη τώρα για το μέλλον. Και μπορώ να τελειώσω για να περάσουμε στις απαντήσεις και ερωτήσεις. Μπορώ να σας πω το εξής τι έλειπε ε, στην Ευρώπη και τι χρειαζόμαστε τώρα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πολύ ισχυρή εποπτεία της αγοράς. Αυτό χρειαζόμαστε. Αν συγκρίνουμε τις ΙΠΑ με την Ευρώπη, ε, μιλάμε για προδιαγραφές ε, λίγο πολύ ισοδύναμες. Η διαφορά είναι ότι στις ΗΠΑ, εδώ και χρόνια, έχουν μια ξεκαθαρή έντολη στην EPA για να έχουν μια στρατηγική και ένα πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς που δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Τώρα λοιπόν έχουμε έρθει ε, και έχουμε δει την ανάγκη να εφαρμοστεί αυτή η εποπτεία της αγοράς. Αλλά κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι σημαντικό είναι και το πώς θα εφαρμοστούν αυτά. Χρειάζεται δηλαδή μια σαφής πολιτική εντολή σε οποιονδήποτε θα είναι η αρχή η οποία θα ελέγχει τις εκπομπές. Χρειαζόμαστε ικανά άτομα γιατί ξέρετε ότι μπορούμε να λέμε το θέμα αλλά αν δεν είναι κανείς εξαιρετικά ικανός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολος ο κλάδος και ε, μπορεί να χαθεί κανείς εύκολα με όλα αυτά τα οποία θα του λένε οι κατασκευαστές. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξεκάθαρη αρμοδιότητα και διαφάνεια. Οπότε ο μόνος τρόπος είναι και προς τα εκεί πάει η πρόταση Κομισιόν. Υπάρχει ένα φόρουμ ανθρώπων με την, υπό την πρωτοβουλία που θα έχουν τα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα, όχι μόνο ποσοτικές εκθέσεις όπου θα μπορούν να αντιληφθούν το τι πάει στραβά και στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά να καταλήγουμε σε μια ε, λύση. Είτε δεχόμαστε είτε δεν δεχόμαστε κάτι. Αυτό νομίζω κάνει την διαφορά και τέλος και καταλήγω εδώ πέρα θεωρώ πως ε, το Jersey είναι απολύτως κατάλληλο για να παίξει ένα τέτοιο ρόλο γιατί είμαστε έτοιμοι, έχουμε τις αρμοδιότητες και την διεθνή φήμη. Αν λοιπόν αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτήν την λύση, μπορούμε να το εφαρμόσουμε από αύριο. Έτσι. Πολύ κατάτα. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Ντεσάντη για όλα αυτά τα ξεκάθαρα και σαφή που μας είπατε και για τις υποσχέσεις της σαφής επίσης που δώσατε για τη δουλειά μας. Τώρα εγώ θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου όχι τόσο στις νομικές πτυχές των εξαρτημάτων αναστολής αλλά σε αυτό που εγώ ονομάζω παράλογη συμπεριφορά των αυτοκινήτων κατά τα τεστ και ιδίως όταν γίνονται στο δρόμο. Ήδη από το 17 και μετά από το 2007 συγγνώμη διαπιστώσατε ότι υπάρχει παράλογη συμπεριφορά κατά τις δοκιμές ε, σε σχέση με το τι γίνεται στο δρόμο και επίσης αυτό διαπιστώθηκε από εκείνη την ε, επικοινωνία με την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ. Και η Γενική Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις ήταν συναρμόδια να νομοθετήσει. Δεν ήταν. Ε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει κάποιο θέμα. Να είμαι σαφής. Ό,τι κάνουμε, πάντοτε το κάνουμε σε πλήρη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Όπως είπα και πριν επομένως, αρχίσαμε την έρευνα για τις πραγματικές εκπομπές NOx, μια που υπήρχε από την DG Envy τον Αύγουστο του 5 η εντολή ξεκάθαρη. Και το ζητήσαμε με Grow, Envy, κλίμα, με όλες τις γενικές διευθύνσεις, όλες, όλα τα ευρήματα που είχαμε, τα, τους δώσαμε τα αποτελέσματα και τα σχετικά έγγραφα. Άρα και η DG Enterprise θα ήξερε για τις επιχειρήσεις δηλαδή. Δεύτερη ερώτηση, κύριε το κ. το πόσο αργά εξελίχθηκαν οι, οι πραγματικές δοκιμές. Και λέει, η μέθοδος RDE θα πρέπει, να ολοκληρωθεί το 2012, δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια από τότε, το 10, το 10, ελέγχθη αυτό για τις πραγματικές εκπομπές. Και τι πήγε στραβά, γιατί πήρε τόσα χρόνια για να αναπτύξετε ε, αυτές τις ε, δοκιμές των πραγματικών εκπομπών. Γιατί πήρε δύο χρόνια, ότι δηλαδή η, η, η μέθοδος πέμψη είναι η καλύτερη. Πέστε μας δύο λόγια. Μάλιστα. Συμφωνώ και έχετε δίκιο. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στην πραγματικότητα. Όταν αρχίσαμε τον Ιανουάριο του 2011 αυτή τη διαδρομή είχαμε τέσσερις μεθόδους να επιλέξουμε. Θα έπρεπε να επιλεγεί ποια θα υιοθετούσαμε. PEMS, modeling, άλλη μία που ήταν η μέθοδος ε, περίπου της ε, που χρησιμοποιούσαν οι ΙΠΑ και, και, το άλλο που ήταν ο τυχαίος κύκλος, random cycle. Δεν υπήρχε συμφωνία από τους συμμετέχοντες. Μέχρι τον Οκτώβριο του 10. Εννοείται και τη βιομηχανία, λέει και κ. Είναι πάνω από 50%. Πόσο, πόσο το έχουμε, δεν ξέρω αν είναι πάνω από 50% τη βιομηχανία αλλά ήταν οι εκπρόσωποι έγκρισης τύπου, οι μη κυβερνικές οργανώσεις, οι αυτοκινητοβιομήχανοι, η επιτροπή, δεν ξέρω αν ήταν 50%. Οπότε, που ενημερώνουμε συνεχώ την ε, Γενική Διεθνή Περιβάλλοντο. Πήρε πολλού μήνε. Τα κουβεντιάζαμε τα ίδια και τα ίδια σε μια σειρά συναντήσεων. δύσκολα από πλευρά πολιτική. Μα τι πολιτική, μιλάμε για τεχνική επιτροπή, λέει και Εγώ μίλησα σε κάποιου που είχαν λάβει το μέρο τη συζήτηση και μου είπαν ότι ήταν ξεκάθαρο ότι επίτηδε παρέλκει τα πράγματα για η μηχανία. Συμφωνείτε, Δεσάντη. Πολλές συνεδριάσεις, πολλές συζητήσεις. Τα ίδια και τα ίδια συζητούσαμε. Ακόμα και πράγματα τα οποία είχαν ήδη ξεκαθαριστεί και αποφασιστεί. Ναι, αλλά καθυστερούσε και η Επιτροπή. Υπήρχαν πρακτικά. Ναι, υπήρχαν πρακτικά για όλα τα συμπεράσματα από την Επιτροπή. Αλλά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς να συμφωνούν όλοι. Ήμασταν επιστημονικοί, δύσκολη κατάσταση. Και πάλι καλά που τελικά του πείσαμε για τη μεθοδολογία που διαλέξαμε. Όλο στοιχείο αυτό που διαλέξαμε εμεί είναι η πιο ανεξάρτητη ε, τεχνολογία. Δεν εξαρτάται δηλαδή από, ε, από κάποιο, κάποια μεταβλητή, ας πούμε, από, το, από τα οχήμα, του υποχήματος κλπ. Και αλλού, και αλλού για το ίδιο ισχύει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Δησάντη που ήρθε και πάλι ενώπιόν μας για να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Ο κύριος Σούτσα δεν μπορούσε να απαντήσει ένα ερώτημα γιατί δεν ήταν τότε υπεύθυνο στο κύριο κέντρο ερευνών. Εσείς όμως ήσασταν το 2012 εκεί πέρα στο κύριο κέντρο ερευνών και Εμείς θέλαμε, θέλουμε να έχουμε τα πλήρη email από αυτήν την εποχή ε, εδώ δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο κύριος Σούτσα είχε πολιτική εντολή να μην δώσει τα email αυτά στην Επιτροπή. Αυτό πρέπει να το αποδείξει κανείς άμα κάνει μια τέτοια κατηγορία. Ξέρω από την άλλη πλευρά ότι έχετε πάρα πολλά email τα οποία ε, τα οποία μπαίνουν σε κάποιο αρχείο. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχετε εσεί στη διάθεσή σα από τι 13 Απριλίου του 2012, συγκεκριμένο email, το οποίο αναφέρεται στο θέμα των εκπομπών ε, οξυδίων του αζότου, λέει ότι τα οξύδια αυτά που εκπέμπονται εξαρτώνται από την θερμοκρασία του κινητήρα. Αλλά λέει εκεί ότι, αν, ότι όταν ε, γίνεται, ξεκινά ο κινητήρας σε χαμηλή θερμοκρασία, τότε είναι πολύ μεγαλύτερη εκπομπή των οξύδιων. Και επομένω υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι γίνεται cycle beating ή hard cycle beating. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ενιών. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να διευκρινίσουμε το εξή. Τότε, όλοι στον κόσμο <clears throat> δεν ένιωθαν καμία έκπληξη που ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ του πραγματικού κόσμου και του κύκλου δοκιμών. Γιατί ο κύκλος δοκιμών ήταν τελείως ανεπαρκής. Επομένω το cycle beating δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν έκπληξη. Δηλαδή ότι αν βγει κανείς έξω από την περιοχή του κύκλου έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό αυτές οι εκπομπές οξυδίων του αζότου μπορούσαν να εξηγηθούν σε τεχνικό επίπεδο και σε ποιο βαθμό όχι. Γι' αυτό θέλαμε να κάνουμε μετρήσεις πραγματικών εκπομπών. Αλλά από την αρχή, αν θυμάστε, όταν ήρθατε σε επαφή με τον επικεφαλής της ε, Υπηρεσίας Μεταφορών της EPA και ρωτήσατε ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν πήρατε αυτές τις εκθέσεις του κοινού κέντρου έρευνων το 2011, <clears throat> είπε δεν με εκπλήσει γιατί ξέραμε ότι ο κύκλος στην Ευρώπη είναι τελείως ανεπαρκής. Όταν βγείτε από τον κύκλο παίρνετε άλλα αποτελέσματα. Γι' αυτό εμείς ξεκινήσαμε να προσπαθούμε να αναπτύξουμε το ταχύτερο δυνατό ένα πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο κύκλο. Γι' αυτό εμείς εστιάσαμε όλες τις προσπάθειές μας στη διαδικασία δημιουργίας ενός κύκλου σε πραγματικές συνδίκες του RD. Και το γεγονό ότι υπήρχε το cycle beating δεν ήταν καμία έκπληξη για μας. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκίζεκε. Ένα πρόσθετο ερώτημα μετά από αυτά τα οποία είπε και ο κύριο Τέρμες αν βλέπουμε ότι δεν είναι πλήρη τα email που έχουμε. Εσείς από την εποχή που ήσασταν ενεργός, 2012-2013, έχετε κρατήσει τα email σας σε κάποιον διακομιστή, τα έχετε σε αρχείο, μπορεί κανείς να τα διαβάσει ή σβήνουν τα email όπως γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο μετά από έξι μήνες. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα για να ξαναβρούμε όλα αυτά τα email. πρώτα απ' όλα. Δεν είμαι εμπειρογνώμων στην πληροφορική. Αλλά με μεγάλη δυσκολία θα μπορούσα να θυμηθώ τώρα πόσα email είχαν σταλεί εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι μπορούμε να ελέγξουμε και πάλι. Βέβαια, εγώ δεν ήμουν αυτό ο οποίο ήμουν εμπεπλεγμένο σε αυτά. Δεν βλέπω πρόβλημα να δούμε όλη την ανταλλαγή email εκείνη την εποχή μεταξύ του κοινού κέντρου ερευνών και των άλλων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Τώρα δεν είμαι ειδικό στην πληροφορική, τι να σα πω κύριος Ματίν. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο αρχιοθετεί τα email που θεωρούνται σημαντικά και σχετικά. Και έχουμε ένα αυτόματο σύστημα που ε, σβήνει τα email μετά από 6 μήνες. Αν δεν έχετε λοιπόν αρχιοθετήσει ένα email σε φακέλους επειδή το θεωρείτε σημαντικό το χάνετε. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος. Φάντε Κάμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σάντι, ε, είστε παλιός στο κύκλο μας. Σήμερα κάνετε μια φυγή προς τα εμπρός. Έξυπνο. Το ερώτημα είναι τι ρόλο παίξατε εσείς και το Ινστιτούτο σας στην επιλογή μεταξύ βενζίνης και δίζελ. Ακολουθήσατε την βιομηχανία ή είπατε ε, προσέξτε παιδιά παραδείγματο χάρη ε, με τα σωματίδια μήπως να το γυρίσετε στη βενζίνη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο. Ε, μία ερώτηση έχω κυρία Πρόεδρε. Έχετε πέντε λεπτά. Α, ε, ας ακούσω τότε. Okay, so first of all... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Η απόφαση για το προς τα που θα πάμε δεν είναι δικιά μας, δεν είναι της Κομισιόν, δεν είναι του Τζέρσι. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε η επιλογή για δίζελ στην Ευρώπη είχε ήδη γίνει. Γιατί αν θυμάστε το δίζελ θεωρείται μια καλή λύση για την Ευρώπη γιατί υπονοεί ε, κάποια εξοικονόμηση καυσίμου, χαμηλότερη κατανάλωση, οπότε θεωρούσαμε ότι ε, αυτό ήταν μια καλή τεχνολογία για την Ευρώπη και ξέρετε πως το βασικό στην Ευρώπη είναι, είναι και, ήταν, είναι και θα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε δεν ε, θεωρείται κακή λύση επί της αρχής. Το πρόβλημα ξεκίνησε αμέσως μετά γιατί είδαμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του Ντιζέλ. Είδαμε ότι ε, πριν από τα οξύδια του αζότου το πρόβλημα ήταν τα σωματίδια Οπότε εστιάσαμε εκεί. Δεν ε, ήταν ε, ε, η δικιά μας η επιλογή το να ήταν καλύτερη βενζίνη ή το ντίζελ. Γιατί ξέρετε, καμία από τις δύο τεχνολογίες αυτές δεν θα είναι η οριστική λύση. Οπότε θα συνεχίσουμε μέχρι τα ηλεκτρικά οχήματα ή κάποια άλλη πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση να είναι διαθέσιμη. Αλλά όσο χρησιμοποιούνται μπορούμε να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο τα μικροσωματίδια πρώτα απ' όλα και μετά τα οξύδια του αζότου. Και μπορώ να σου πω πως αν χρησιμοποιηθεί σωστά η τεχνολογία, το ντίζελ έχει τον αντίκτυπο τον ίδιο με τη βενζίνη. Ίσως και καλύτερο αν σκεφτεί κανείς ε, το DGTI. Αλλά από την περιβαλλοντική σκοπιά με τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν τώρα στην εξάτμιση του δίζελ είναι καλύτερο. Ε, θεωρείτε πως έχετε εξετάσει επαρκώς επιστημονικά τα πιθανά μειονεκτήματα του δίζελ. Ναι, νομίζω ότι πάντα δημοσιεύαμε όλα τα αποτελέσματα που βρήκαμε. Είχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Ε, Έχουμε υπογράψει και συνεργασία με όλα τα επιστημονικά κέντρα, ερευνητές ε, στον κόσμο. Έχουμε μνημόνια με Κίνα, Ιαπωνία, Κορία, Κορέα, Ηνωμένε Πολιτείες. Το έχουμε δει από όλες τις πλευρές το ζήτημα. Και πώς ε, βλέπετε το πώς διάλεξε τα αποτελέσματα της η Κομισιόν. Δηλαδή ε, κάνατε δοκιμές, βρήκατε κάποια ασυνέπεια, ήταν για σας ικανοποιητική η αντίδραση στα ευρήματα αυτά. Όχι. Ε, πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να γίνει μια διάκριση. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα εδώ. Η μία δουλειά είναι να βελτιώσουμε την γνώση για να βασιστεί εκεί η μελλοντική νομοθεσία. Αυτή είναι η έρευνα που κάνουμε. Ε, άλλη δουλειά είναι η έγκριση τύπου, είναι άλλη δουλειά δηλαδή. Κάποιος κοιτάει προς τα μπρος και κάποιος κοιτάει προς τα πίσω και αστυνομεύει. Οπότε όσον αφορά το μέλλον, την έρευνα, την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, αν έρθετε να μας δείτε στην Ίσπρα θα δείτε εκεί πέρα τα πρώτα φίλτρα σωματιδίων που αναπτύξαμε εμείς ε, μαζί με τη βιομηχανία. Τώρα το... η διαδικασία αυτή δοκιμών πραγματικού δρόμου, αυτή την αναπτύξαμε εμείς πάλι θα χρησιμοποιείται παγκοσμίω. Οπότε έρευνα, στήριξη της καινοτομίας, ναι, αυτό κάνουμε ως επιστήμονες, ερευνητές. Όσον αφορά την έγκριση τύπου, ε, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Και αυτό ακριβώς λείπει. Ε, κρίμα, κρίμα για σας. Όπως είπα και πριν, ε, αυτό λείπει στην Ευρώπη. Αν αποφασίσουμε να έχουμε ένα σύστημα σοβαρό, αξιόπιστο, με διαφάνεια για να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα, μόνο αυτό το κομμάτι λείπει. Η εποπτεία της αγοράς να βρεθεί μια αρχή η οποία θα έχει την αρμοδιότητα και την ε, μεθοδολογία να τα εφαρμόσει αυτά σωστά. Τότε η Ευρώπη θα είναι πρώτη παγκοσμίω. Ε, κύριε Μπονεφά. Καλημέρα κύριε Δεσάντη. Αν επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Σούτσα, το 70% του ρόλου σας είναι η καλή εφαρμογή της νομοθεσίας των ευρωπαϊκών κανόνων και ιδίω του κανονισμού του 2007. Και 30% πράγματι είναι η έρευνα νέων τεχνολογιών που θα είναι πιο αποτελεσματικές. Μέσα σε αυτό το 70% όμως, μήπως θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι είναι μια γενική εντολή να εξασφαλίσετε ότι τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες και οι ρυθμίσεις. Δεν είναι αυτό μια γενική εντολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών, γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί την καλή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όχι, μαντάμ, όχι, λέει ο κύριος Ντισάντη. Το να υποστηρίξουμε την νομοθεσία σημαίνει να φέρουμε επιστημονικά στοιχεία και να τα δώσουμε στους λήπτες αποφάσεων. Είτε είναι Ευρωπαίοι, είτε είναι εθνικά κράτη κτλ και μετά να δούμε κατά πόσο αυτοί οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν. Αλλά η επιβολή της νομοθεσίας δεν είναι στην εντολή μας. Και τι ακόμα λείπει. Αν μας είχαν ζητήσει να πάρουμε στοιχεία από τους κατασκευαστές ή από τις αρχές έγκρισης τύπου θα το είχαμε κάνει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν ενεπλάκημεν καθόλου στην εποπτεία της αγοράς αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε ακόμα η εποπτεία της αγοράς. Γιατί αυτό έχει μείνει στην <clears throat> αρμοδιότητα κάποιων των κρατών μέλων. Κάποια το πράττουν, κάποια όχι. Εμείς όχι. Μα ξέρατε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, λέει η κυρία. Είχατε αυτό το, τη γνώση του προβλήματος γιατί προχωρήσατε προς την τεχνολογία μετρήσεως σε πραγματικές συνθήκες τον Οκτώβριο του 2015 μετά από την υπόθεση Volkswagen είναι σαφές ότι είχε ζητηθεί από το κοινό κέντρο ερευνών να δει με τα κράτη-μέλη τι ξέρανε για τις ε, συσκευές αυτές της διατάξης αναστολής. Αυτό ήταν πράγματι σαφές στο έγγραφό σας. Είχατε λοιπόν μια έντολη. Τον Οκτώβριο του 2015 ήσασταν ακόμα αρμόδιος. Τι έγινε λοιπόν με την μελέτη αυτή, με την έρευνα αυτή, για την οποία πήρατε εντολή να δείτε τι γίνεται με τα, από τα κράτη-μέλη για τις ε, διατάξεις αναστολής. Αν κατάλαβα καλά, αναφέρεστε στο πιο πρόσφατο τεστ, αυτό που είναι πριν από φέτος. Αναφέρομαι σε αυτό το έγγραφο το οποίο διάβασα, δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε αλλά μας δόθηκε να το διαβάσουμε. Οκτώβριος του 2015 είναι τα πρακτικά της συνεδρίασης. Όταν ξέρω το σκάνδαλο, ζητήθηκε από το κέντρο να μελετήσει με τα κρατημέλη ε, σε όλα τα κρατημέλη όπου υπήρχε τέτοιο εξάρτημα και να γίνει μια τέτοια παρουσίαση του τι μπορεί να γίνει με, για αυτές τα, τα εξαρτήματα. Οπότε είχατε όλα τα στοιχεία, είχατε και την εντολία. Yes. Yes, we... Α, μάλιστα. Και μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, Μέσα μας εργαζόμαστε με την DigiGrow και τις ε, αρχές σύγκρισης τύπου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει, να συντονιστούμε. Να βοηθήσουμε ούτως ώστε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες για αυτά τα τέστα να τελείω διαφορετικά στα κράτη-μέλη. Οπότε δώσαμε τι κινητήριε γραμμέ που ακολουθήθηκαν από τα εθνικά ε, προγράμματα. Το κάνουμε αυτό αμέσω. Και επίση από την ε, Γενική Διεύθυνση Grow το Μάιο φέτο την εντολή του να αρχίσουμε να κάνουμε εμεί οι ίδιοι μια εποπτεία της αγοράς. Τέσσερα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και το Σεπτέμβριο γνωστοποίησαμε το αποτελέσμα στην ε, Γενική Διεύθυνση Grow και λίγες μέρες μετά σε εσά από ό,τι ξέρω. Άρα υπάρχει η σχετική έκθεση από όσο ξέρω. Όχι από ό,τι ξέρω. Αφού λέτε όμως ότι είναι προσβάσιμη θα τη δούμε. Χτες είχαμε μία συνάντηση στην Επιτροπή και μας είπαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο έκθεσης το οποίο έχει σταλεί στη Γενική Διεύθυνση Grow. Τέσσερις δοκιμές, Euro 6 και τα αποτελέσματα σας έχουν διαβαστεί. Δεν ξέρω, μπορεί να τα πάρετε αύριο, σήμερα. Μάλλον σήμερα, μάλλον σήμερα λέει ο Πρόεδρος. Στις 7 η ώρα. Στις 7 λέει ο κ. Ντεσάντη. Mr. Gerbrandi. Gerbrandi. Α, εγώ πάλι. Αν θέλετε. Έχετε ζήσει το λόγο, λέει εδώ πέρα η λίστα. Κύριε Μάισνερ, ευχαριστούμε κύριε Ντεσάντη που ήρθατε. Είπατε επιλέξει ότι αναπτύσσουμε τα καλύτερα τεστ, καλύτερη τεχνολογία, καλό αυτό για μας. Και είπατε επίση ότι η υποπτία τη αγορά είναι πολύ σημαντική. Αλλά θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να προσπαθήσουμε περισσότερο. Είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίω. Τώρα, πότε το πρώτο σκεφτήκατε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνετε τέτοιου είδου εποπτεία τη αγορά. Πότε σα προέκυψε για πρώτη φορά αυτή η ιδέα, πότε το προτείνετε στην Κομισιόν αυτό σαν ιδέα όταν αρχίσαμε να συντάσσουμε με τους ανθρώπους της DigiGrow ε, την πρότασή μας για τη νέα έγκριση τύπου. Άρα ούτε το 9 ούτε το 10, αλλά πιο πρόσφατα. Α, καλώς. Πρώτη μου ερώτηση ήταν αυτή, λέει μέσα. Ε, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Είπατε να αναπτύξαμε την καλύτερη τεχνολογία για τεστ. Για πέστε μας. Νομίζετε ότι ακόμα δεν είναι δυνατόν να κλέψουν οι αυτοκινητοβιομήχανοι σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές. Γιατί σκοπό είναι να μην μπορούν να κλέψουν στο μέλλον. Θεωρείται ότι η τεχνολογία όμως είναι τέτοια που μπορεί να κρύψει ή τέλο πάντων μπορεί η τεχνολογία να αποτρέψει κάποιου από να χρησιμοποιούν τέτοιου μηχανισμού διάταξη αναστολή. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό λέει ο Παραλαμβάνω. Το, το, το είναι το καλύτερο διάρμο που θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερη βελτίωση. Και αυτό είναι κάτι που θα υιοθετηθεί παγκοσμίω. Όμω, πάντοτε ο διάβολο κρύβεται στην εφαρμογή. Οπότε, εάν δεν υπάρχει μια αρμόδια αρχή που να εφαρμόσει αυτό, τότε δεν θα υπάρξει καμία εγγύηση. Δεν υπάρχει ποτέ εγγύηση απόλυτη. Άρα να έχει την εντολή κάποια αρχή που να μπορεί να εξετάσει τι κάνει αυτή την μηχανία, τι γίνεται με την έγκριση τύπου, όταν υπάρχει υποψία, επομένω μόνο έτσι. Άρα εμεί του δώσαμε το καλύτερο δυνατό μέσο. Όμω θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με έξυπνο τρόπο. Και μην ξεχνάτε ότι η μεθοδολογία για τις πραγματικές ακόμα δεν έχει θεσπιστεί. Το έχουμε στην έγκριση τύπου, αλλά για την ε, εποπτεία της αγοράς ακόμα δεν έχει μπει στη δέσμη μέτρων. Γι' αυτό σας λέω, εκεί πέρα είναι το, το κλειδί, η υλοποίηση να υπάρξει κάποιο οργανισμό οργανισμός και αυτοί να εφαρμόσουν την μεθοδολογία μας. Ναι. Είπατε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε κατά πόσον κάνουν τη δουλειά του τα κράτη-μέλη και αρμόδιε αρχές. Γιατί όχι. Δεν μπορούσατε να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει. Υπήρχε η νομοθεσία. Εσείς είσαστε ο σύμβουλος της Κομισιόν. Αφού δεν ήσασταν ικανοποιημένοι με τα πράγματα, είπατε τίποτα στην Κομισιόν. Τους είπατε να ελέγξουν περισσότερο τα κράτη-μέλη ή δεν μπορέσατε. Και πάλι είχαμε πολλές συζητήσεις <clears throat> με τους συναδέλφους μας. Μα ούτε ένα email από όλα αυτά δεν υπάρχει. Τίποτα δεν έχει διασωθεί, λέει ο 7 η ώρα το βράδυ. Θα σας τα στείλουμε, λέει ο κύριος Δησάντη. Όχι. Υπήρξαν συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο, υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το πώς να αναπτύξουμε με τον ταχύτερο τρόπο τη λύση. Αυτό ήταν ο κύριος στόχος μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι όταν ξεκινήσετε από το μηδέν γιατί δεν υπάρχει ακόμα η νομική βάση και δυνατότητα. Λειτουργήσαμε λοιπόν επί τη βάση της εντολής μας που ήταν να λύσουμε το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατό και με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μα δεν έγινε. Γιατί θεωρήσατε ότι τα πράγματα είχαν επιληθεί και μετά ξαναρχίσανε να συζητούνται πάλι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ο οποίος φταίει για όλα αυτά. Έχουμε 28 κράτη-μέλη, επομένως δεν είναι εύκολο να πούμε ότι φταίει κάποιος. Αυτό είναι αποτέλεσμα του κατακαιρματισμού του ευρωπαϊκού συστήματος. Υπάρχουν πολλά κράτη, πολλές απόψεις. Πρέπει να ζήσουμε λοιπόν με αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται στα κρατη λέει η κυρία Μάσινα. Είναι πολύπλοκο το σύστημα. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνένεση. Δεν έχουμε μία αρχή όπως οι ΗΠΑ στην Αμερική, η οποία αποφασίζει τέρμα. Εμείς πρέπει να πείσουμε μέσω των επιτροπών τα κάτι μέλη να υπάρξει μια ομοφωνία ή έστω μια πλειοψηφία. Και κατά δική μου άποψη δεν είναι το καλύτερο. Από θα μπορούσατε να έχετε κάτι σαν την EPA. Αυτό σημαντικό ερώτημα, αλλά βλέποντας την κατάσταση τώρα στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα όνειρο και μόνο. Γιατί έχετε τις εθνικές αρχές έγκριση τύπου σε κάθε χώρα. για να τις συγκεντρώσετε όλες αυτές σε μόνο μία <clears throat> αρχή είναι πολύ δύσκολο. Πιο λογικό θα ήταν να υπάρξει αυτό που γίνεται η πρόταση της Κομισιόν, να υπάρχει ένα φόρουμ που θα υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων. Αλλά η ανταλλαγή δεδομένων ακόμα δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχετε μία συνένεση όταν υπάρχουν διαφωνίες και κάποιος να έχει την εξουσία να φέρει τα πράγματα σε ένα αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε απλώς ε, ένα κοινό κέντρο ερευνών που χρηματοδοτείται με όχι φυσική αλλά με πολύ λίγα χρήματα. Τούρμες. Σάντι, με κάθε σεβασμό, όταν λέτε ότι έχουμε την πρώτη και τη δεύτερη δουλειά, υπήρχε μια τρίτη δουλειά που είχατε. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάζει εάν οι εγκρίσει τύπου, αν οι αρχές που κάνουν τις τύπου κάνουν σωστά τη ε, δουλειά τους. Και ο κύριος Ποτότσνικ, ο επίτροπο, ο κύριο Φάλκενμπεργκ, ε, ο Γενικός Διευθυντής ε, Περιβάλλοντος, η νομική υπηρεσία της Διεύθυνσης περιβάλλοντο είπαν πως υπήρχε βάση για διαδικασία παράβασης και άρα θέλουμε να μάθουμε ποιος ήταν επικεφαλής της ομάδας σας το 2010, ποιοι ήταν οι εταίροι σας ε, στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, ποιος συνέταξε την έκθεση. Αυτά. Αυτά είναι εύκολα. Εγώ ήμουν επικεφαλής με τμήματάρχη τον Καζιμίρ. Η συντάκτες έκθεση είναι Πιέρ Μπονέλ, Μάρτιν Βάις και άλλοι. Εύκολα μπορούμε να το βρούμε. Οι συνομιλητέ μας επίσης γνωστοί. Χρησιμοποιήσατε email. Όχι. Κύριε Τούρμες, ε, προσωπικά όχι, γιατί ε, ε, ο διευθυντής δεν αντάλλασε email. Μα στο επιχειρησιακό επίπεδο. Δηλαδή έχετε κόσμο στην Ίσπρα, στις Βρυξέλλες, πώς επικοινωνούν. Με email, με τι. Κοιτάξτε και πάλι... Ναι, ναι μάλλον ναι. Ε, δεν είναι περίεργο. Μεταξύ τη γενική διεύθυνση ε, ε, Επιχειρήσεων Κλίματος, ριβάλλοντο και ημών να υπάρχει αλληλογραφία. Οπότε και εσείς είστε έκπληκτό προφανώς που δεν υπάρχει ούτε ένα email για την Επιτροπή μα. Δεύτερον, Είπατε κάτι πριν για τις ΕΠΑ. Είπατε πως η διαδικασία δοκιμών και η νομική βάση στις ΕΠΑ δεν διαφέρει τόσο πολύ από την Ευρώπη. Μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν τόσο μεγάλη διαφορά όσο μας λέει η αυτοκινητοβιομηχανία και κάποιοι λομπίστες. Δεν είναι θέμα νομοθεσίας. Ε, όχι, όχι, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο πλευρά προδιαγραφών πολλά πράγματα είναι ίδια. Το ζήτημα των διατάξεων αναστολής είναι ίδια. Έχουμε 300.000 κινητήρες δίζελ στη ΣΥΠΑ και το ανακάλυψαν εκεί. Εμείς έχουμε εκατομμύρια δίζελ, κινητήρες δίζελ στην Ευρώπη και δεν το βρήκαμε. Πού οφείλεται αυτό. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι στην εποπτεία της αγοράς. Γιατί και, δεν το ανακάλυψε η EPA αυτό. Με όλες τις δοκιμές που έκαναν. Δεν το ανακάλυψαν γιατί το λογισμικό που καταλάβαινε ότι το αυτοκίνητο περνούσε τεστ ε, μπορεί να υπάρχει μια άλλη διαφορά. Ότι είναι ε, αρχή περιβάλλοντος στις ΗΠΑ ενώ στην Ευρώπη είναι αρχή βιομηχανίας. Αυτή είναι η, διαφορά. Είναι διαφορά. Όπως σας είπα είναι η εποπτεία της αγοράς Εσεί θα αποφασίσετε πολιτικά. Εγώ ως τεχνικό μπορώ να πω ότι η εποπτεία τη αγορά είναι για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Δεν θα ήταν πιο λογικό να είναι στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αντί για επιχειρήσεων. Και επί την ευκαιρία το κέντρο σας είχε συμβόλαιο με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος από τα 2007 το 2005 και το 2007 ξαφνικά δεν είναι αρμοδιότητα της γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και πήγε στη Γενική Διεύθυνση ε, Επιχειρήσεων. Γιατί. Κύριε Τούρμε, μη ρωτάτε εμένα γιατί ένα χαρτοφυλάκιο πήγε από τη μια Γενική Διεύθυνση Κομισιών σε άλλη. Μα ε, δεν σα εξέπληξε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν ήταν πια αρμοδιότητα της γενική διεύθυνση περιβάλλοντο, αλλά πήγανε στην βιομηχανία. Δεν σα εξέπληξε. Εξέπληξε, αλλά εφόσον συνεχίζαμε τις δοκιμές και όπως πριν για μένα δεν υπήρχε πρόβλημα. Βεβαίως ε, θα ήθελα να πω συνήθως ε, στην Κομισιόν δεν είναι μία γενική διεύθυνση αρμόδια, εμπλέκονται κι άλλες. τελευταία ερώτηση για τις φορητές συσκευέ. Αυτές για τα γεωταχή αναπτύχθηκαν από το 2007 και μετά. Γιατί χάσαμε δύο χρόνια το 11 και 12. Το Πολυτεχνείο του Γκράτς ε, που πλήρωνε η αυτοκινητοβιομηχανία ε, είχε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργιστεί, καθυστερούσαν, τι έκαναν. Και γιατί η Γενική Διεύθυνση ε, Επιχειρήσεων που προέτρεπε συνεδριάσει δεν επέμενε ότι τέρμα τα αντίφραγκα. Κοιτάξτε, τώρα είναι εύκολο να ασκούμε κριτική εκ των υστέρων, αλλά πιστέψτε με, ε, αναπτύσσαμε μια νέα τεχνολογία, εντελώ νέα και έπρεπε να υπάρχει συνένεση μεταξύ των ειδικών. Οι ειδικοί έχουν άποψη, ε, έχει ο καθένας ε, την δικιά τους, τη δικιά του εμπειρογνωμοσύνη. Εμείς το κέντρο μας κάναμε πολλές δοκιμές για να βρούμε τα υπέρ και τα κατά για κάθε μεθοδολογία. Μάλιστα, το, το τελευταίο που θέλω να σας πω. Αλλά τελευταίο λέει η πρόεδρος ποιος ήταν υπεύθυνο για τις δοκιμές στο κέντρο σας, ποιος ήταν ο ομολογός σας στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και χρειαζόμαστε τα email. Ναι, ναι, θυμάμαι τους δύο βασικούς από τη δικιά μας την πλευρά ήταν ο Μάρτιν Βάις και ο Πιέρ Μπονέλ. Αυτοί ήταν οι δύο για εμάς, δεν κάνω λάθος. Και στην άλλη πλευρά, ο Φιλίπ Ζαν Στάνιγκερ. Ε, εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Να το διασταυρώσουμε, λέει Και τελευταία ερώτηση από την κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Τεσσανή. Για πέστε για τον ε, driving cycle. Το ξαναείπαμε, αλλά νομίζω θα πρέπει να το ξανααναφέρουμε. έχουμε τον κανονισμό 715 και λέει εκεί ότι αυτός ο driving cycle δεν ε, εκπροσωπεί πλέον τις ε, πραγματικές ε, συνθήκες. Αυτά το 2007 πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αν σιγά σιγά να καταλήξετε στο RD σαν στρατηγική και σαν μέθοδο. Βεβαίω και ήταν δύσκολο να την τελειοποιήσετε, να την ολοκληρώσετε και να φτιάξετε σε κάτι ακριβές και αξιόπιστο, αλλά όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο τεστ όπως το Artemis δηλαδή Cycle κλπ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το χρησιμοποιεί για το διοξείδιο του αζότου, το είπε πέρσι. και αλλού επομένως χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος. Το PEMS είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι εύχριστο. <coughs> Γιατί επομένως δεν φροντίσετε να υπάρχει κάποιο άλλο τεστ. Όχι, όχι στα, στα αγγλικά θα σα τα πω, όχι στα ιταλικά. Να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Το PEMS συμπληρώνει το driving cycle. Άρα και τα δύο χρειάζονται. Το PEMS χρειάζεται μόνο για τις εκπομπές εκτός κύκλου. Δεν θα χαιρετίζαμε χρόνο με το Artemis γιατί ήταν ένας κύκλος ίσως υπερβολικά δυναμικός. Θα πρέπει να περάσουμε μια διαδικασία ελέγχου για την ανεπαραγωγημότητα. Ε, θα, θα έπαιρνε τουλάχιστον δύο χρόνια. Ακριβώς το χρόνο που χρειαστήκαμε για να αναπτύξουμε αυτόν τον κύκλο που χρησιμοποιεί παντού στον κόσμο. Άρα καλύτερα έτσι. Γιατί το Άρτεμις ξεκίνησε από το δεδομένο που πήραμε από Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Τώρα μπορεί να έχουμε στοιχεία από παντού. Άρα ήταν ε, πολύ καινοτόμα αυτή η προσπάθεια. Να έχουμε αυτό το drivable δυναμικό τεστ. Άρα δεν θα ωφελούσε το Άρδενης, ακόμα και αν ήταν ε, δυναμικό. Άλλο σκοπό είχε για ανάλυση των εκπομπών και όχι για ε, έγκριση τύπου. Επομένως, κατεβλήθη προσπάθεια στα πλαίσια του ΟΗΕ, είχαμε αυτό το νέο δυναμικό τεστ και τελικά αυτό ήταν η σωστή επιλογή, γιατί θα βαζόταν σε δεδομένα από παντού, από όλο τον κόσμο. Και το RD επομένω είναι το σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα, που είμαι σίγουρος ότι ελήφθη η σωστή απόφαση. Εντάξει, τώρα ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω, είπαμε και πριν. Έτσι είναι το ισχύον σύστημα. Πρέπει και σε τεχνικό επίπεδο να υπάρχει συμφωνία και συνένεση. ευχαριστώ για την απάντηση. Αλλά παρά το ότι υπήρχαν όλες αυτές οι τεχνικές δυσκολίες για την εφαρμογή των μεθοδολογιών τεστ, νομίζω ότι αυτά τα δύο χρόνια για τα οποία μιλήσατε, πόσο είπατε να κερδίσουμε χρόνο όμως ήταν και θέμα ανθρωπίνων ζώων το πόσο κόστησε αυτός ο χρόνος. Γιατί σίγουρα και υπήρχαν επιπτώσεις από τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, από το οξύδιο του αζότου, ε, στο πόσοι πέθανε. Μιλάμε για πρόωρους θανάτους 70.000 ετησίω. Άρα παράλληλα με την ανάπτυξη του αντί θα μπορούσατε να εξετάσετε το αν υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ θα λίγα, το πρόβλημα δεν ήταν ο κύκλος. Έπρεπε να γίνει αντικατάσταση με πιο δυναμικό κύκλο, ήταν οι εκπομπέ εκτός κύκλου. Οπότε αυτές δεν μπορούσαμε να τις πάρουμε. Μόνο με το δυναμικό κύκλο που είναι μια βελτίωση. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τα προβλήματα όλων των εκπομπών κύκλου. Γι' αυτό είπαμε ότι επικεντρωθήκαμε στο RD και το νέο δυναμικό τεστ στα πλαίσια του ΟΗΕ. Ε, ναι, αλλά η ίδια η Ιταλική υπηρεσία που το αυτά και το Άρτεμις λέει για κάποια αποτελέσματα, κάποιου είδου τιμές, κάποια διαφορά μεταξύ των 5 και των 7 φορών. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα της ρήπανσης. Ε, θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η μεθοδολογία. Όχι. Δεν θα έκανε διαφορά. Τώρα έχουμε δύο, δύο μεθόδους. Έχουμε την ε, άρτεμη με από και την άλλη το παγκόσμιο τεστ. LLDP. Άρα από πλευρά δυναμικού κύκλου θεωρώ ότι έχει κλείσει η ιστορία. Ευχαριστώ. Έτσι έχουμε κλείσει τις δύο ακροάσεις. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε τα ερωτήματα που κάνετε τις δηλώσεις. Θα υπάρξουν και κάποια πρόσθετα γραπτά ερωτήματα που θα σας αποσταλούν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν και αν έρθουν τα email αργότερα μπορούμε να έχουμε κάποια ευκαμψία για τις ερωτήσεις και ζητώ από όλους από την Κομισιόν να μας βοηθήσουν να έχουμε αυτά τα email. Η επόμενη μας συνεδρία είναι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Καλό Σαββατοκύριακο.